So, ladies and gentlemen, please take your place. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε αμέσως. Τρεις η ώρα. Good, meine Damen und Herren, damit eröffne ich wieder die Sitzung. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Μοσχείου Όπως ξέρετε αναμεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίασή μας και θα ξεκινήσουμε αμέσως με την ημερήσια διάταξη το σημείο 7, το οποίο δεν προλάβαμε το πρωί να το συζητήσουμε. Πρόκειται για το πρωτόκολλο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών της και της Κορέας. Και βεβαίως αυτό γίνεται για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ο εισηγητής ε, με μία ταχεία διαδικασία θα μας παρουσιάσει. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί ε, συζήτηση και αντιρρήσεις. Ε, θα δώσω βεβαίως ε, το λόγο αμέσως στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα είπατε περίπου όλα όσα έπρεπε να λεχθούν. Δεν πρόκειται για ένα θέμα επίμαχο είναι ένα τυπικό θέμα, αν θέλετε, διότι πρέπει απλώς να προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση μετά την προσχώρηση της Κροατίας. Όπως ξέρετε αυτή η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Κορέα έγινε μετά την, ε, το, την Λισαβόνα και ε, το Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του και μετά όταν τον Ιούλιο 2013 προσχώρησε η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε προσωρινή εφαρμογή. Τώρα θα πρέπει λοιπόν να επισημοποιήσουμε την κατάσταση και το πρόσθετο πρωτόκολλο με το οποίο η Κροατία προσχωρεί σε αυτήν την συμφωνία και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την συγκατάθεσή του ε, που την έδωσε τον Μάρτιο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, τις ευρωεκλογές. Το μόνο που σας ζητώ και σας συνιστώ αγαπητοί συνάδελφοι, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτό το πρωτόκολλο, ούτω ώστε η Κροατία να γίνει ε, πλήρες μέλος από την άποψη αυτή. Αυτά μπορώ να πω. Είμαι σύντομος, διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν είναι επίμαχο. στην σκιώδη γιατί θα δώσω το λόγο, εάν θέλετε βεβαίως, δεν είναι υποχρεωτικό δεν βλέπω όμως ε, σκιώδεις εισηγητές ή εισηγήτριες. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Η Επιτροπή... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα πρωτόκολλα που αφορούν την προσαρμογή μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών στην προσχώρηση ενός νέου κράτους όπως την Κροατία. Είναι κάτι το οποίο έχει δημοσιευθεί, θα αρχίσει να ισχύει με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουνίου του 2013 καθότι όλοι οι εμπλεκόμενοι από την Κροατία φορείς θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα αυτής της συμφωνίας και αυτού του πρωτοκόλλου, καθώς και αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της αναδρομικής ισχύω έχει γίνει και σε άλλες φορές. Έχουμε προχωρήσει βεβαίω στην ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, είναι όμως απαραίτητη και η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ε, ο εισηγητής, να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί στηρίζετε τις προτάσεις μας και εγώ απλώς επανέρχομαι στις αρχικές μου συστάσεις. Πρόεδρος, 5 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή δηλαδή, είναι η, προ... η την υποβολή τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι το σημείο που αφορά το 10, 11, 12 και 13. Πρόκειται δηλαδή για τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία, τη Μόλδομα και τη Γεωργία. Μέχρι το 13 δηλαδή, 11, 12, 11 και 12. Όπως είχα πει και σήμερα το πρωί, πρόκειται όσον αφορά το πρώτο σημείο, δηλαδή την συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία, ε, για ένα θέμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο πρέπει να διεκπαιρεώσουμε με ταχύτητα. Θέλουμε να επισπεύσουμε δηλαδή λίγο τη διαδικασία. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Από την άλλη, όπως ξέρετε, ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν έτσι ώστε η κύρωση να γίνει από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ταυτόχρονα με αυτή που θα γίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη δηλαδή ολομέλεια στο Στρασβούργο να ψηφίσουμε για την συμφωνία αυτή. Πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία η οποία δεν είναι η κανονική μας διαδικασία. Είναι μια πολύ πιο ταχεία διαδικασία. Μπορούμε λοιπόν με μια επιστολή να συγκεκριμενοποιήσουμε την θέση μας, τη γνωμοδότησή μας. Θα συμφωνήσουμε εδώ επί της ουσίας και ο Acting Deputy Director General, ο Ιγνάσιο Ντεσέρο, από την Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εδώ και βεβαίως θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτής της Συμφωνίας Σύνδεσης αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε στη διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών μας με χώρες της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Όπως ε, πολύ σωστά είπατε, στην περίπτωση της Ουκρανίας είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε παράλληλη ε, επικύρωση από το Ουκρανικό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι ο πρόεδρος Ποροσέγκο έχει την πρόθεση να γίνει η κύρωση μέσα στο Σεπτέμβριο. Όπως ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία διμερών διαβουλεύσεων. Με... Έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και την ε, Ουκρανία για να δοθεί απάντηση σε διάφορα ζητήματα που έφυξε η Ρωσική Ομοσπονδία. Έχουμε μία ε, αποστολή του Επιτρόπου Ντεκούτ ε, στις 12 ε, Σεπτεμβρίου στην Ουκρανία και θα εμπλακούμε επικοδομητικά σε αυτές τις συζητήσεις περνώντας ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρεί κανεί ότι η συμφωνία μα αυτή με την Ουκρανία θα δημιουργήσει προβλήματα για την ρωσική οικονομία. Για κάποια κανονιστικά θέματα υπάρχει ευελιξία στη συμφωνία και θα πρέπει να ε, διευκρινίσουμε προς την Ουκρανία και τη Ρωσική Ομοσπονδία ότι τα στοιχεία αυτά ευελιξία υπάρχουν ακριβώς για αυτό το σκοπό, ούτως ώστε η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας να προχωρήσει με ομαλό τρόπο. Ε, φυσικά είναι ε, σημαντικό το πολιτικό μήνυμα που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα βήματα που θα κάνουμε για να δείξουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο για την επικύρωση θα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Επίσης, ευχαρίστω να δεχτούμε οποιασδήποτε ερωτήσεις θα έχουν τα μέλη της Επιτροπής μας, ε, εδώ, της Επιτροπής εδώ, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τις άλλες χώρες όπως, ε, όπου εφαρμόστηκαν προσωρινά οι συμφωνίες αυτές. Ξέρετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Ρωσική Ομοσπονδία έλαβε κάποια περιοριστικά μέτρα απέναντι στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα για την Μολδαβία, όπου η Ρωσία εφαρμόζει όχι μόνο ε, απαγόρευση 60% των ε, εξαγωγών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά ε, έχει ε, έπαιρνε εισαγάγει και δασμούς αντίθετα με την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και η Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση να δώσουμε ένα μήνυμα υποστήριξης προς τους ε, Μολδαβούς ε, φίλους μας και, για, και εντελώς σε προσωρινή ε, βάση να λάβουμε ειδικά μέτρα ευελιξίας για εξαγωγή προς εμάς των προϊόντων που δεν μπορούν να εξαχθούν προς την Ρωσία. Ευχαρίστω να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις έχετε, αλλά προς το παρόν ε, υποθέτω ότι θα θέλετε να εστιάσετε τη συζήτηση ε, το θέμα της Ουκρανίας και χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να προχωρήσει παράλληλα με την Ουκρανία στην ε, κύρωση αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε τις πολιτικές ομάδες. Καταρχήν, ε, πρώτη σε δύναμη, το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, από ό,τι καταλαβαίνω, πρόκειται για ένα πολιτικά λεπτό θέμα. Υπάρχει ανάγκη να πίεση χρόνου, να επισπεύσουμε τη διαδικασία και την κύρωση αυτή τη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες. Την ίδια ώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι όντως όλα τα πρακτικά θέματα επιταχύνονται και την ίδια ώρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εάν λοιπόν είναι δυνατόν ακριβώς επειδή είναι λεπτό το θέμα να μην είμαστε ιδιαίτερα αν θέλετε, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοιτώντα ποιε θα μπορούσαν να είναι τυχόν ε, δευτερεύουσες επιπτώσεις, επιπτώσεις σε άλλες συμφωνίες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα ένα τμήμα της Ουκρανίας, και το λέω αυτό με ήπιο τρόπο, είναι υπό τον έλεγχο ε, μιας άλλης χώρας. Με ποιο τρόπο λοιπόν εμείς μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο ήπιες, ευέλικτες διατάξεις για κάποιους οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν. Ας ξεκινήσουμε με την κύρωση, ας μην βεβαίως επιβραδύνουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά ξέρω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μην δημιουργήσουμε αρνητικές επιπτώσεις ε, σε αυτή τη συμφωνία. Ποιος άλλος θέλει το λόγο από τους σοσιαλιστές. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε με ε, την διπλή επικύρωση της συμφωνίας και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της γεωπολιτικής δραματικής κατάστασης που γνωρίζουμε όλοι. Θα ήθελα επίσης να έχω μερικές πρόσθετες πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά ε, με αυτήν την θετική αλλά κάπως ενηγματική ε, πρωτοβουλία από την Ουκρανία τον Απρίλιο, εάν η Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει μια αξιολόγηση της κατάστασης ε, σχετικά με τις προτεραιότητες, με το πλαίσιο και αν υπάρχουν ε, διευκολύνσεις ε, εμπορικές, θέματα τελωνιακά και σε σχέση με την Κρυμαία θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις εισρωές αγαθών κλπ. Ε, αν έχει γίνει ήδη από την ειδική ομάδα, αν έχουν ε, γίνει εργασίες σχετικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συντηρητικοί μεταρρυθμιστές. Sorry, Emma will be with us. Με ε, συγχωρείτε. θα ήθελα να θέσω σχετικά με το θέμα της Ουκρανίας με απασχολεί το στρατιωτικό θέμα ε, στην Συμφωνία Σύνδεσης και τι ε, ε, σημαίνει αυτό σε σχέση με την όλη γεωπολιτική κατάσταση μου φαίνεται ότι πηγαίνει πέραν της εμπορικής συμφωνίας και είναι κάτι το πολιτικό. Διαρωτώ με εάν οι όροι αυτοί είναι ήπιοι, θα γίνουν πιο σκληροί αλλά αυτό που με απασχολεί και πάλι και με ανησυχεί, το είπα εδώ στην Επιτροπή Εμπορίου, ίσως, ίσως μπαίνουμε πολύ στο πολιτικό πεδίο ε, ασχολούμεθα με τις θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις, με την βοήθεια ε, στην οικονομία. Είναι πολιτικά αυτά τα θέματα με την Ουκρανία και οι συνέπειες ε, σε σχέση με τα πολιτικά, με την άμυνα θα είναι τραγικές ίσως. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την σαφή παρουσίαση των εισηγητή. Κατανοούμε και υποστηρίζουμε ε, το ότι είναι κατεπίγουσα η ε, επικύρωση λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων ε, που έχουμε ως προς την ασφάλεια και ως γενικά επειδή υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Το βασικό θέμα είναι να υπάρξει μια διατηρήσιμη, ε, βιώσιμη πολιτική ε, λύση. Οι κυρώσεις δεν ξέρω αν ε, θα διανοίξουν το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ νομίζω ότι η Συμφωνία Σύνδεσης έχει γίνει το σύμβολο, ένα σύμβολο ευρωπαϊκού προσανατολισμού για τους Ουκρανούς πολίτες στην Πολωνία και στην Ουκρανία ε, πριν από 25 ε, χρόνια το κατακεφαλήν εισόδημα ήταν ε, σήμερα στην Ουκρανία είναι 7.000 και στην Πολωνία 20.000. Βλέπετε 2,5 φορές περισσότερο δυνατή η οικονομία της Πολωνίας ενώ ήταν στο ίδιο επίπεδο πριν από 25 χρόνια βλέπουμε τι γίνεται όταν υπάρχουν ατομικές ελευθερίες και γι' αυτό η Συμφωνία Σύνδεσης έγινε σύμβολο και τόσο σημαντικό θέμα. Υποστηρίζουμε λοιπόν την ταχύρυθμη ε, διαδικασία και την επικύρωση στην επόμενη σύνοδο του Στρασβούργου ή δυνατόν αυτής της Συμφωνίας Σύνδεσης και των Συμφωνιών Ελευθέρων Συνελλαγών. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα στην Επιτροπή σε σχέση με τη συμφωνία της διαπραγματεύσεις και τις συνέπειες. Πρώτον, ε, σχετικά με τις ε, τριμερείς ε, συνομιλίες Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρανία, Ρωσική Ομοσπονδία και ίσως Δυτική Ένωση, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιες είναι οι δυσκολίες. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, μπορείτε να μας υπενθυμίσετε την ασυμματρία του Συμφωνία Σύνδεσης ε, σε σχέση ε, με την πρόσβαση στην αρχή ε, πώς θα είναι για την Ουκρανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα. Ευχαριστώ, Ιγκούε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Εξεπλάγεν όταν είπε στην αρχή ότι χρειαζόμαστε μία πολύ ταχεία διαδικασία. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν ε, αυτή η διαδικασία κύρωσης, ναι ή όχι, θέλουμε να προχωρήσουμε αυτόν τον τρόπο. Έχω την εντύπωση ότι δεν τηρούμε τις δημοκρατικές ε, διαδικασίες και τις εγγύσεις. Τι να σας πω, οι ευρωπαϊκές εκλογές έγιναν πριν από λίγο καιρό και αυτά πρέπει να τα προσέχουμε γιατί ξέρετε τα προβλήματα που δημιουργούμε με τέτοιες ε, διαδικασίες. Υπάρχει μελέτη αντικτύπου όσον αφορά παραδείγματος χάρη κάποιες ελλείψεις όπως αυτόν τον πολύ σημαντικό στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα, τι σημαίνει για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν χωρίς κανέναν έλεγχο προχωρήσουμε στην κύρωση αυτής της συμφωνίας με αυτήν την ταχεία διαδικασία. Εδώ στην Επιτροπή, αν θυμάστε, με τον, Επιτροπή, με τον ε, εισηγητή της Επιτροπής μας, τον κύριο Παρεύσκη, είχαμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλες αυτές οι ε, επιπτώσεις και μάλιστα είχαμε πει ότι θα γίνει και ε, μία μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση για όλες τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Εδώ λοιπόν εγώ αναρωτιέμαι όλα αυτά τα θέματα έχουν απαντηθεί. Δηλαδή η κύρωση αυτής της συμφωνίας με αυτήν την επισφευμένη διαδικασία είναι κάτι που σε αυτήν την καυτή κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία θα βοηθήσει. Μήπως, μήπως με έναν άλλο τρόπο θα είχαμε βοηθήσει πολύ πιο θετικά. Τρίτη ερώτηση που θέλω να κάνω, που αφορά επίσης αυτή τη συμφωνία, υπήρχε και το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ερωτώ λοιπόν, την Επιτροπή. Αυτό ίσως δεν έχει άμεση σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά έχει σχέση με τη συμφωνία. Τι κάνουμε για να καταπολεμήσουμε τη διαφορά, γνωρίζοντας πως έχει σήμερα η οικονομική και η πολιτική κατάσταση της Ουκρανίας. Τελειώνοντας, έχω άλλη μια ερώτηση. Ξέρετε ότι έχει γίνει η, μια μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιους πολύ συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικούς στόχους. Αναρωτιέμαι λοιπόν στην Ανατολική Ουκρανία τι μπορούμε πολύ συγκεκριμένα να κάνουμε για να βοηθήσουμε να μην υπάρξει μετατόπιση πληθυσμών, κάτι που σιγά σιγά γίνεται και αλλαγή των, ε, της σύστασης ε, των κατοίκων, των πολιτών που ζουν σε αυτή την περιοχή. Καθότι σήμερα επικρατεί μια νέα, πολύ ενισχυτική κατάσταση στην περιοχή αυτή και θέλουμε να ξέρουμε αν μπορούμε κάτι να κάνουμε για να το εμποδίσουμε. Οι πράσινοι δεν ζητούν το λόγο. αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δεν ε, συμφωνώ συχνά με τον κύριο Σούλτς όπως ξέρουν τα μέλη της ε, Επιτροπής, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί του εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία σύνδεσης πάρα πολύ αμφιλεγόμενη, πάρα πολύ πολιτική, που θα έχει επιπτώσεις και συνέπειες που χρειάζεται να τη σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά και δεν υπάρχει κανένα σημείο ότι ο κύριος Ρόντερ ότι τα έχει σκεφτεί καν όλα αυτά και η πρόταση που έχουμε στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Δεν καταλαβαίνω τι, δεν ξέρω τι έχετε καπνίσει, κάτι που θα έμεινε από τη δεκαετία του 60 ίσως, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι εντελώς αλόκοτη αυτή η προσέγγιση η στιγμή είναι κατάλληλη για πάρα πολύ προσεκτικό προβληματισμό, πολύ προσεκτική σκέψη όλων των συνεπειών, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα ε, εθνικά κράτη της ε, Ευρώπης, για τις χώρες μας, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τις οικονομίες μας και δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι οποιοδήποτε έχει σκεφτεί οτιδήποτε από όλα αυτά, ότι τα έχει ε, μετρήσει ε, όλα αυτά, παρά μόνο ότι ε, έχουμε τον Αμερικάνο πρέσβη. Και ας προχωρήσουμε κι εμείς μαζί με τους Αμερικάνους και σε μία ακόμα συμφωνία σύνδεσης. Παρεπιπτόντως, υπάρχουν πολλοί στο Κοινοβούλιο που διαφωνούν σε βάθος για αυτά που λέτε εσείς και ο πρώην επιτροπός σας. Όσον αφορά αυτά τα ποσά που είπατε για το ΑΕΠ της Ουκρανίας και της Πολωνίας, 7.000. 7.000. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν κρέμομαι από το στόμα σας. Ε, εντάξει, 7.000. Αλλά θα δεχτείτε ότι ένας από τους λόγους που η Πολωνία τα πήγε τόσο καλά ήταν λόγω των μαζικών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν η Ουκρανία γινόταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα περίμενε και θα έπαιρνε σύντομα ε, τεράστιες επιδοτήσεις. Και η δική μου ψηφοφόρη, η ψηφοφόρη του κυρίου Μάρτιν και ίσως όχι η δική σας αλλά και πολλών άλλων ψηφοφόροι ε, σε αυτή τη φάση μας ζητάνε περικοπές. Δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό όλο αυτό και απλώς δείχνει την ε, ουτοπία την, ε, στην οποία ζείτε. Και ελπίζω ότι τα παράλογα αυτά σχόλιά σας θα διορθωθούν και τέλος, κάτι ακόμα ήθελα να πω. Προφανώς ανησυχούμε πάρα πολύ για την Ουκρανία, για τα 70 εκατομμύρια. 58. 45 λοιπόν περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Ανησυχούμε για αυτούς. Και θα θέλαμε τα μέτρα ελέγχου της μετανάστευσης που υπάρχουν να παραμείνουν σε ισχύ και δεν θέλουμε με οποιαδήποτε συμφωνία να ανοίξει πίσω πόρτα για την κατάργηση των θεωρήσεων ή των διαβατηρίων. Είχα κάτι να πω και για, την, για τις προτάσεις που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις τριμερείς σχέσεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο καταστροφικό, αλλά δεν είναι αυτό θέμα αυτής της Επιτροπής μας. Θέλω λοιπόν ε, από τον κύριο Μπερσέρο ε, κάποιες ε, πιο σοβαρές απαντήσεις. Λοτόφσκι. Dziękuję Σας ευχαριστώ. Από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ αναφερόμαστε στην υποστήριξη της ε, Ουκρανίας, ενώ διαδραμαζείται πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Βεβαίως είμαστε υπέρ της Ουκρανίας, θέλουμε να την υποστηρίξουμε, ενώ βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Σαν ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή, τι μπορούμε να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Η προκειμένη κατάσταση μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι αφενός η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος, από την άλλη συνεχίζουμε να τους προμηθεύουμε με όπλα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να συνεχίζουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές με τη Ρωσία. Ποιο άλλο θέλει να πάρει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον Ιγνάσιο. Θα σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένος στις απαντήσεις μου, όσο μπορώ απαντώντας σε ερωτήσεις που έγιναν. Πρώτη ερώτηση. Οι συνέπειες του που συμβαίνει για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να προμηθεύσει οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά και μέχρι τώρα παρέχουμε ένα προτιμησιακό καθεστώς στην Ουκρανία. Αυτό που θέλουμε είναι να θεσμοθετηθεί μια πάγια πρακτική όσον αφορά αυτό το προτιμησιακό καθεστώς και για πρώτη φορά θα ανοίξει η αγορά της χώρας αυτής ε, με ειδικού όρους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες Ευρωπαϊκή Ένωσης, με την εφαρμογή κανόνων και ρυθμίσεων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βεβαίω υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε ε, διατάξεις για τις εμπορικές αυτές συναλλαγές και ένα τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου φυσικά θα πρέπει να υιοθετηθεί από την Ουκρανία. Έχουμε δημιουργήσει μία task force, μία ειδική ομάδα εργασίας. Η... Τα μέλη αυτής της task force σήμερα δεν είναι εδώ, αλλά στο μέλλον με μεγάλη χαρά θα έρθουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της Επιτροπής σας. Έχουμε στηρίξει λοιπόν την Ουκρανία, τις αρχές της Ουκρανίας, στις βασικές τους πολιτικές επιλογές έτσι ώστε προοδευτικά και σταδιακά να ευθυγραμμιστούν και να υιοθετήσουν τις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προχωρήσαμε στις διμερείς μας ε, συνομιλίες και θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής σας να κατανοήσουν ότι αυτές οι διμερείς ε, συνομιλίες έχουν ε, προχωρήσει σημαντικά. Η Ρωσική Ομοσπονδία βεβαίως ανησυχεί και έχει εκφράσει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας σύνδεσης. Εμείς θεωρούμε ότι τα επιχειρήματά τους δεν ευσταθούν Έχουμε ξεκινήσει παρόλα αυτά ένα διάλογο, καθότι ο διάλογος με την Ουκρανία συνεχίζεται και σκοπός μας είναι να υπάρξουν κάποιες εγγύησεις, κάποιες διασφαλίσεις, έτσι ώστε να μην ανησυχεί η Ρωσική Ομοσπονδία εξαιτία αυτής της συμφωνίας. Αυτές είναι οι διμερείς συνομιλίες, τις οποίες έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούλιο και θέλουμε να διασφαλίσουμε την ε, υλοποίηση αυτής της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών χωρίς να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ρωσική οικονομία. Η κύρωση αυτής της συμφωνίας είναι μια πολιτική επιλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς θα αποφασίσετε, εάν ναι ή όχι, θέλετε να δώσετε αυτό το μήνυμα στην ε, Ουκρανία η οποία πραγματικά έχει υιοθετήσει μια πάρα πολύ θαραλέα στάση να προχωρήσει και να ευθυγραμμιστεί με τις ε, δικές μας ρυθμίσεις και κανονισμούς. Βεβαίως για οποιαδήποτε επιπλέον ερώτηση μπορείτε να μας την απευθύνετε και με μεγάλη χαρά θα σας ε, απαντήσουμε και θα σας δώσουμε ή δίποτε πληροφορία που αφορά αυτήν την συμφωνία σύνδεσης. Το θέμα της ασυμμετρίας που υπάρχει σε αυτήν την συμφωνία. Υπήρξε μια ερώτηση για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σιγά σιγά ανοίξει την αγορά της στην Ουκρανία και με την συμφωνία αυτή η αγορά της Ουκρανίας σταδιακά τα επόμενα 3-5 χρόνια, 7 χρόνια θα ανοίξει για κάποια ειδικά προϊόντα και τομείς προβλέπεται μια ακόμα μεγαλύτερη χρονική περίοδος για το άνοιγμα της ουκρανικής αγοράς, όπως παραδείγματο χάρη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θεωρούμε όμως ότι σε γενικές γραμμές αυτή η συμφωνία είναι θετική και για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την ουκρανική οικονομία και προβλέπει και επιβάλλει στην Ουκρανία κάποιες μεταρρυθμίσεις οικονομικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται λοιπόν να υποστηρίξει την εργασία και τις συνομιλίες που έχει ξεκινήσει διμερώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια αυτής της ειδικής ομάδας εργασίας της Task Force. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος άλλος θα ήθελε να κάνει ερώτηση, να δευτερολογήσει. Ο Χέλμουτ. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Θα είμαι πιο συγκεκριμένος στην ερώτησή μου. Ποιες επιπτώσεις βλέπετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οικονομία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοιτώντας αυτές τις προθεσμίες που περιέχει αυτή η συμφωνία. Ερωτώ για τα δημητριακά, για τα γεωργικά προϊόντα. Ξέρουμε πολύ καλά τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ουκρανίας και Μοντσάντο για τα δημητριακά και δεν μπορούν αυτά τα προϊόντα να φτάσουν και να έχουν πρόσβαση στην δική μας αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον τομέα της ενέργειας, επανέρχομαι. Αν κοιτάξετε τα άρθρα της συμφωνίας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας χωρίς να έχουμε εκτιμήσει, αξιολογήσει τις πραγματικές επιπτώσεις για την οικονομία μας. Αυτό το κάνουμε σε όλες τις συμφωνίες. Συνήθως συζητούμε επί δύο χρόνια, αξιολογούμε και εκτιμούμε τις επιπτώσεις. Είναι περίπλοκα τα θέματα αυτά, είναι επίμαχα. Και πραγματικά δεν είμαι καθόλου ήσυχος. Δεν κάνω τις ερωτήσεις αυτές πραγματικά για να σας εμποδίσω, αλλά θεωρώ ότι αν θέλουμε να έχουμε μία θετική συνεισφορά δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέζουμε για συμφωνίες οι οποίες επηρεάζουν και τυχόν με αρνητικό τρόπο μπορεί να επηρεάσουν πολύ ευαίσθητους τομείς όπως αυτό των δημητριακών, των γεωργικών προϊόντων, της ενέργειας κτλ. Ερωτώ λοιπόν, έχουμε κάποια εκτίμηση αυτών των επιπτώσεων. Έχει κάνει κάτι η Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνω ότι η σιωπή έχει επίσης κάποιο νόημα. Αλλά έχω παρόλα αυτά μια ερώτηση, παρόλο που δεν έλαβα απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση μου. Ξεχάσατε να μου απαντήσετε ή δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Euh, Καλημέρα. Ε, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εδώ, ίσως δεν έχει πολλά να κάνει σχετικά με την Διατλαντική Συμφωνία, είναι καλό θέμα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για τις ε, συζητήσεις με την Ουκρανία και την Ρωσία, την κατάσταση των διαπραγματεύσεων βεβαίως. Ίσως στο επόμενο θέμα θα ασχοληθούμε ε, με την κατάσταση, αλλά μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η ατμόσφαιρα, ποια είναι η θέση της Ρωσίας σε σχέση με το θέμα αυτό. Για να έχει κανείς μια πλήρη εικόνα της ε, συμμετοχής ε, της Ευρώπης ε, στην σταθεροποίηση και στην ανάπτυξη της Ουκρανίας θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η εκτίμηση, τρέχουσα εκτίμηση της Επιτροπής ως προς το πόσο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει για αυτήν την σταθεροποίηση. Από ό,τι θυμάμαι είναι 10-15% των ε, συνολικών αναγκών, 15 δισεκατομμύρια περίπου. Οπότε 1,5 δις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ίσως και 10. Αυτό είναι σημαντικό ακόμα πιο σημαντικό διότι με τη Συμφωνία Σύνταξης και την Εμπορική Συμφωνία και Συμφωνία Πρόσβασης στην Αγορά θα έχει η Ουκρανία μέσα να ωφεληθεί για την οικονομική της ε, ανάπτυξη. Αυτό είναι τελικά πιο σημαντικό. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση. Υπάρχουν διατάξεις στη Συμφωνία Σύνδεσης ή θα μπορούσαν να υπάρχουν διατάξεις στην Συμφωνία Σύνδεσης ε, που θα, ε, θα χαλαρώσουν, ε, θα διευκολύνουν το καθεστώς των θεωρήσεων. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις που αφορούν την συμφωνία με την Μολδαβία, το προτιμησιακό καθεστώς, τις επιπτώσεις, τις κυρώσεις προς τη Ρωσία και αυτά που συμβαίνουν σήμερα και πλήττουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς τις αποφάσεις που πήρε η Ρωσία. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και να απαντηθούν στα πλαίσια της ίδιας συζήτησης. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις αλλά αν ξέχασα κάποια από αυτές, μην διστάσετε παρακαλώ να μου την υπενθυμίσετε. Πρώτον, οι ερωτήσεις του κυρίου Τσόσερ σχετικά με την ενέργεια και τη γεωργία. Πρώτον, ελπίζω να είναι ε, κατανοητό σαφέστατα ότι σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμφωνεί σε καμία απολύτως αλλαγή για το STS, για την γεωργία. Νομίζω ότι αναφέρεται τα, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. οργανισμούς. Η ε, Ουκρανία συμφώνησε σταδιακά να ευθυγραμμίσει την νομοθεσία της STS με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το κάνει σταδιακά και μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας θα μας πει ποιες είναι οι προθέσεις της σχετικά με αυτή τη ε, ε, σταδιακή ευθυγράμμιση της νομοθεσίας θέματα STS, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλάξει οτιδήποτε ε, όσον αφορά την νομοθεσία για τα θέματα SPS. Φυσικά δεν μπορεί να έχει κανείς μια συμφωνία αν δεν, αν δεν κάνει παραχωρήσεις αλλά είπαμε ότι αυτές οι παραχωρήσεις δεν θα έχουν καμία σημαντική αρνητική συνέπεια για την ευρωπαϊκή αγορά. Και να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση μονομερός εφαρμόζει κάποιες ε, παραχωρήσεις προς την Ουκρανία και οι συνέπειες αυτής της συμφωνίας θα είναι ότι ε, από την άλλη μεριά και η Ουκρανία σταδιακά θα ανοίξει τη δική της αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για την ενέργεια. Οι ενεργειακές διατάξεις για τη συμφωνία αυτή και πάλι ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι αντικατοπτρίζουν μία δέσμευση εκ μέρους της Ουκρανίας που έχουμε γιατί ήδη συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας να ευθυγραμμίσουν σταδιακά την νομοθεσία τους και στο θέμα της ενέργειας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω ε, εν δυνάμει τι συνέπειες θα έχει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας και δεν μπορώ να ε, κάνω υποθέσεις για το τι θα κάνουν τρίτες χώρες, τι δεν θα κάνουν. Αλλά υπάρχουν ειδικέ διατάξεις ώστε η Ουκρανία να εξασφαλίσει την ε, διέλευση, το τρανζιτ. Για τις τριμερείς τώρα συνομιλίες θα είμαι πάρα πολύ σαφής θα απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Γιαντό. Όντω, την περασμένη Δευτέρα συμμετείχα στι εργασίε των τριμερών διαβουλεύσεων με την Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία. Ήταν μια πολύ καλή αντιπροσωπεία, πολύ υψηλού επίπεδου και εκ μέρου των δύο κυβερνήσεων και νομίζω ότι έγινε μια επικοδομητική και επαγγελματική συζήτηση. Εμείς προχωρήσαμε σε πολύ λεπτομερείς επεξηγήσεις, παραδείγματο χάρη όσον αφορά τις διατάξεις της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, γιατί είμαστε ευέλικτοι και πώς είμαστε ευέλικτοι, πώς θα δώσουμε στην ε, Ουκρανία το ελεύθερο να αποφασίσουν αυτή το ρυθμό ευθυγράμμισής τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένας ε, ε, λόγος η Ρωσία να φοβάται ότι θα πληγούν οι εξαγωγές της προς την Ουκρανία διότι θα εγκαταλειφθούν τα παλιά πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται στην Ουκρανία. Ε, είναι επικοδομητική η ατμόσφαιρα λοιπόν των συζητήσεων. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε. Θα συμμετάσχει η Κομισιόν και στο Μίνσκ, γιατί έχουμε προσκληθεί και στις 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο όπου ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καθησυχάσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία ότι δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται τη συμφωνία αυτή αλλά ότι αντίθετα θα συνεργαστούμε πολύ στενά μαζί τους για να παρακολουθήσουμε την ε, εφαρμογή, την υλοποίηση της ε, συμφωνίας αυτής με τρόπο που θα καθησυχάζει οποιαδήποτε θεμητή ανησυχία τους. Και ελπίζουμε πραγματικά πάρα πολύ ότι η Ρωσική ε, Ομοσπονδία δεν θα κάνει στην Ουκρανία αυτά που έκανε με τη Μολδαβία, γιατί ξέρετε ότι με τη Μολδαβία υπήρχε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ε, και όπως με τις χώρες ΚΑΤ και η Ρωσική Ομοσπονδία αποφάσισε να αναστείλει την συμφωνία αυτή για ένα πολύ μεγάλο μέρος του εμπορίου της με την Μολδαβία. Ελπίζουμε ότι με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν θα λάβει την ίδια θέση η Ρωσική Ομοσπονδία απέναντι στην Ουκρανία. Τώρα, όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία, δεν εκπροσωπώ την ε, Task Force για την Ουκρανία ακριβώς, αλλά η ε, από ό,τι ξέρω, ήδη έχει 600, 600 εκατομμύρια συν 250 εκατομμύρια κινητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 100 εκατομμύρια κατά τους προσεχείς μήνες ε, σε δάνεια και επιχορηγήσεις αντίστοιχα. Ε, και αυτό θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και έχουμε καθήκον και ευθύνη να παρέχουμε την μέγιστη δυνατή υποστήριξη για την οικονομική ανάκαμψη της ε, χώρας και για να ε, το υποστηρίξουμε αυτό. Ακούστηκε η ερώτηση σε ποιο βαθμό εμπορικά θέματα θα αποτελέσουν αντικείμενο της υποστήριξης. Μα όλα αυτά που λέμε έχουν να κάνουν και με εμπορικά θέματα, με προσαρμογή των κανονισμών και των προτύπων τους προς τα ευρωπαϊκά ε, στάνταρ. Το ίδιο και για τα τελωνία. Υπάρχει μια πολύ σαφής επιλογή εκ μέρους της Ουκρανίας να κινηθεί προς ε, αυτή την κατεύθυνση και εμείς είμαστε πρόθυμοι να ε, δώσουμε αυτή την υποστήριξη που χρειάζονται. Φοβάμαι ότι δεν είμαι εξοικειωμένος με θέματα θεωρήσεων, ε, αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με την FTA, με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για τις υπηρεσίες, αλλά τίποτα για τις θεωρήσεις. Αν ε, θέλετε μπορώ να ρωτήσω τους συναδέλφους μου και να ενημερώσω την Επιτροπή σας. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα στην FTA σχετικά με τις θεωρήσεις. Ενώ ε, στις γενικότερες διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης, ειλικρινά δεν ξέρω τι ε, ισχύει. Ε, άκουσα όμως τις ερωτήσεις σας και ευχαρίστως να προσπαθήσω να βρω την απάντηση. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε προηγουμένως για την Κρυμαία. Τι γίνεται με την Κρυμαία. Ξέρετε ότι δεν έχουμε δεχτεί την ε, προσάρτηση της Κρυμαίας από την Ρωσική Ομοσπονδία και γι' αυτό έχουμε λάβει διάφορα μέτρα στη σχέση μας με την Κρυμαία. Αλλά αυτό είναι μάλλον πολιτικό θέμα και όχι εμπορικό. Τέλος, δεν θέλω να πω τίποτα για τις ρωσικές κυρώσεις. Ξέρουμε τι μέτρα πήραν τον Ιούλιο. Η Κομισιόν βεβαίως ε, πήρε μέτρα για την υποστήριξη των παραγωγών μας για να ε, αντισταθμιστεί αυτή η εντελώς άδικη ε, ενέργεια. Το θέμα ε, το έχουμε πάει και στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αυτό δεν είναι σημερινό θέμα σήμερα, αλλά δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αντιπίνων, μια σου και, μια σου και μία μου, ε, το βρίσκουμε πολύ λυπηρό ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πήρε αυτά τα μέτρα. Ε, εμείς πήραμε μέτρα για να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς μας και σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να φέρουμε, δεν έχουμε φέρει, το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να φέρουμε αυτό το θέμα ενώπιον του ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον να θέλει άλλη συμπληρωματική ερώτηση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το θέμα αυτό. για τα τέσσερα αυτά σημεία. Δεν άκουσα κάποιον να είναι εντελώς αντίθετος με την συμφωνία μεταξύ των δύο προέδρων όσον αφορά αυτήν την ταχεία διαδικασία που θα λάβει χώρα παράλληλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Γι' αυτό και θα στείλω μια επιστολή στην Επιτροπή ΑΦΕΤ στον Πρόεδρο, στην οποία θα ε, ξεκαθαρίσω ποιες είναι οι δικές μας θέσεις. Θα αναφερθώ στο θέμα της παρακολούθησης της υλοποίησης αυτής της συμφωνίας και θα αναφέρω ιδιαίτερα και το θέμα του αντικτύπου των επιπτώσεων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ουκρανία. Επίσης, θα αναφέρω ρητά ότι αυτή η διαδικασία είναι κάτι που δικαιολογείται αποκλειστικά και μόνο από τις ε, έκτακτες συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν την ε, ε, περιοχή και ότι δεν μας επιτρέπει, όπως κάνουμε συνήθως, να αξιολογήσουμε τις συνέπειες μιας τέτοιας σημαντικής οικονομικής συμφωνίας. Ο Χέλμουτ. Η δική μου όμως θέση δεν ήταν αυτή. Εγώ είπα ότι διαφωνώ με το πώς προχωράμε και θα ήθελα όλες οι πολιτικές ομάδες να πάρουν θέση και να εκφραστούν για το πώς τοποθετούνται σε σχέση με αυτήν την ταχεία διαδικασία. Οι άλλες πολιτικές ομάδες, λέει ο Πρόεδρος, θέλουν να σχολιάσουν περαιτέρω το θέμα αυτό. Η κυρία Λεπέν. Δεν μπορείτε επειδή, να πείτε ότι επειδή δεν θέτουμε ερωτήσεις συμφωνούμε με αυτή τη διαδικασία. Ορισμένες ερωτήσεις τέθηκαν. Εγώ προσωπικά οι πολλαπλοί βουλευτές που εκπροσωπώ σε αυτήν την Επιτροπή είναι τελείως αντίθετοι με την διαδικασία που προτίθεστε να εφαρμόσετε. Λάμπστορφ. Και εγώ θα ήθελα εδώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως και με τον συνάδελφο Σόλτς, με την συνάδελφο Λεπέν. Βλέπω εξάλλου ότι συμφωνούν πολύ μεταξύ τους, πλήρη συμφωνία. Εμείς οι φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι είναι μια πολύ άτυπη διαδικασία, άτυπη όσον αφορά ε, την συνήθη διαδικασία. Πρόκειται όμως, αν θέλετε, και για μια πάρα πολύ άτυπη και έκτακτη κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι δεν ε, σταματάμε μπροστά σε μια χείρα βοηθείας την οποία ξεκινήσαμε να τίνουμε προς την Ουκρανία. Συμφωνώ απολύκτως με τον Γράφον Νάπερς. Αυτή η διαδικασία δεν είναι συνήθις, σίγουρα αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι και η κατάσταση δεν είναι συνήθις. Αν ε, είχαμε έναν ε, συνήθι τρόπο να την αντιμετωπίσουμε, ουσιαστικά θα παίρναμε τη στάση, θα υιοθετούσαμε τη στάση που υιοθετούν όλοι αυτοί που είναι κατά αυτής της βοήθειας. Και αυτό βεβαίως εδώ θα δημιουργήσει ένα τεράστιο χάσμα. Ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι αντίθετοι και δεν θέλουν να κάνουμε καμία ούτε πολιτική, ούτε οικονομική, ούτε ανθρωπιστική κίνηση. Αλλά για αυτές τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν εκεί, η Ουκρανία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και θα πρέπει να το καταλάβετε. Πρέπει να καταλάβετε όλοι εσείς που ζήσατε παρόμοιες συνθήκες ότι πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και πρέπει να κινηθούμε. πάρα πολύ σύντομα. Δεν έχουμε αντίρρηση στην διαδικασία, αλλά οι λόγοι, τα επιχειρήματα υπάρχουν. Όταν, όταν θα παραπέμψουμε το θέμα στην ΑΦΕΤ και στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία είναι έκτακτη, αλλά επίσης ε, έχουμε μια ε, θέση ε, που δεν είναι συνηθισμένη στην Ουκρανία, σύνηθη κατάσταση. Είχαμε εκλογές, νέο κοινοβούλιο, νέες περιστάσεις μέσα σε αυτήν την μοναδικό πλαίσιο των καταστάσεων. Δεν πρέπει να αντιτεθούμε στη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιτιθέμεθα σε αυτήν την ταχύρυθμη διαδικασία. Υπάρχουν πολύ λεπτά μέτρα, ευαίσθητα μέτρα. Η ανάπτυξη διαλόγου, συνεργασίας μεταξύ για το, το θέμα της ασφάλειας ε, και της άμυνας σχετικά με την ακαιρεότητα των ε, συνόρων νομίζω βρισκόμαστε σε πάρα πολύ λεπτή, βίφοβη, ε, ε, επικίνδυνη κατάσταση, κυρίως ως προς τις σχέσεις ε, ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία και θα στείλουμε ένα πολύ κακό μήνυμα στη Ρωσία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ λεπτά και ευαίσθητα, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι. Κύριε Βεβαίως συμμερίζουμε ε, τα όσα είπε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση ως προς την διαδικασία. Θεωρούμε ότι βεβαίως δεν είναι κλασική η κατάσταση. Σε μια κλασική περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοια διαδικασία, αλλά τα σημάδια τα πολιτικά είναι διαφορετικά εδώ και τα μηνύματα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ επίμαχη. Υπάρχει εδώ διχογνωμία εδώ στο Κοινοβούλιο όπως και στην Ουκρανία. Νομίζω θα έπρεπε να το αναβάλουμε το θέμα αυτό λόγω ε, της διαφωνίας και να μην πάμε να ψηφίσουμε. Η αναβολή δεν είναι κάτι που μπορούμε να το επιλέξουμε γιατί αυτό δεν έχει ληφθεί σαν απόφαση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορετικές θέσεις που εκφράστηκαν. Οι πολιτικές ομάδες εκφράστηκαν ξεχωριστά, η πλειοψηφία εκφράστηκε υπέρ. Όπως λοιπόν είπα, θα στείλω στον κύριο Μπροκ, πρόεδρο της Επιτροπής ΑΦΕΤ και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, θα στείλουμε μία επιστολή εκφράζοντας πολύ συγκεκριμένα τις αντιθέσεις και τις επικρίσεις που ακούστηκαν και εκφράστηκαν εδώ, κατά πρώτο λόγο, και δεύτερον, ότι θεωρούμε αυτή τη διαδικασία μια εξαιρετική και μη κανονική διαδικασία, η οποία δικαιολογείται λόγω των έκτακτων συνθήκων, και τρίτον, θα αναφερθούμε βεβαίως και στην έλλειψη αξιολόγησης αντικτύπου όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Ένα διαδικαστικό που αφορά τον κύριο Μάρτιν. Δεν κατάλαβα ποια είναι η θέση των σοσιαλιστών. Είστε υπέρ ή απλώς ε, δηλώσατε ότι θα απέχετε. Δεν ξέρω, θα ήθελα να ξέρω. Ποια είναι η θέση των ε, σοσιαλιστών, γιατί μιλήσατε για πλειοψηφία της Επιτροπής. Μπορούμε να ψηφίσουμε, σας παρακαλώ. Ζητώ ψηφοφορία. Από τη στιγμή που ζητάτε ψηφοφορία, θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ της ε, προτινόμενης διαδικασίας. So, one.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 Είναι σαφής η πλειοψηφία υπέρ. Εξού και θα κάνουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Σε τρία λεπτά θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ελέγξτε παρακαλώ ότι έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Ευχαριστώ. Νομίζω δεν με είδατε, Πρόεδρε. Θεωρώ πραγματικά ότι πρόκειται για μία εντελώς άτυπη διαδικασία και με αυτήν την σύντομη ψηφοφορία βεβαίως βλέπετε την πλειοψηφία με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι αντικειμενικός. Λοιπόν, σε δύο λεπτά ψηφίζουμε. Έχουμε την κανονική μας ψηφοφορία. Herr Ober. Okay, four o'clock. We know that we vote first on the we vote first on the amendment. Uh, first this one. First this one, right? Yeah, yeah, yeah. And then the amendment. Okay. Liebe Kollegen. Συνάδελφοι, ελπίζω να έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ψηφοφορίας και θα ξεκινήσουμε Θα ξεκινήσουμε με τον προϋπολογισμό. Υπάρχει συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 της κυρίας Κέλλερ. Όχι, καταπίπτει. Κατόπιν έχουμε την 5 της κυρίας Κέλλερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 της κυρίας Μακλάκιν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προχωράμε στην τροπολογία 7 κυρία Σάκε. Σε δύο τμήματα ψηφίζουμε. Το πρώτο τμήμα καταρχήν ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 8 της κυρίας Μακλάκιν. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 του κυρίου Μπέγκε του εισηγητή ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά ξαναψηφίζουμε την τροπολογία 9 Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Ένας παραπάνω. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 του κυρίου Μάρτιν. Ποιος είναι υπέρ. κατά, ελέγχουμε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας για τη 10. Ένας παραπάνω από την ομάδα των συντηρητικών. Ψήφισε. Τέλος. Εγκρίνεται η τροπολογία 10. Περνάμε στην 11 της κυρία Σάκε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 11. Τροπολογία 12 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 του κυρίου Σόλτς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Αρχή. Τέλος. Απορρίπτεται. Γιάννη, καμφισβήτησες την ε, εκτίμησή μου. Τελειώσαμε με την ψηφοφορία των τροπολογιών. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα θα ψηφίσουμε τις γραμμές του προϋπολογισμού με εισηγητή πάλι τον ε, Ράινερ Μπέγκε. Ψηφίζουμε τώρα τη γραμμή 20.01.01.01. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ε, τροπολογία της κυρίας Σάρκε για συμπλήρωση του 0202 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατόπιν πρόταση του κυρίου Σόλτ για την γραμμή 0204 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία για την γραμμή 2102-77-29 της κυρίας Αρένα. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος αρχή της ψηφοφορίας τέλος απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε για το συνολικό κείμενο για να διαπιστώσουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε αυτή τη φορά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνονται οι τροποποίησεις αυτές. Συγχαρητήρια κύριε Μπάγκε. Ολοκληρώσαμε και την ψηφοφορία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται τα περιβαλλοντικά αγαθά στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει διμερείς προτάσεις, συζητήσεις και έχει υποβάλει προτάσεις και θεωρώ ότι είναι και ενδιαφέρον αλλά και απαραίτητο να ακούσουμε για το πόσο έχουν προχωρήσει αυτές οι συνομιλίες και να δούμε πώς ε, συμβαδίζουν με άλλες ε, διαπραγματεύσεις ε, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μεταξύ της 5ης Ιουνίου και της 31ης Ιουλίου συνεχίστηκαν αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες και θα πρέπει να δούμε εδώ αυτός ο πρώτος γύρος που έλαβε χώρα 9 και 10 Ιουλίου πώς ε, προχώρησε. Ο δεύτερος γύρος θα λάβει χώρα το φθινόπερο. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κεντρικό θέμα για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε και ένα άλλο θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχει ένα ξεχωριστό σημείο που αφορά τη Ρωσία. Εσείς στα συνοπτικά σας σχόλια είπατε ότι καλύψαμε όλα τα σημεία και τη Μολδαβία και τη Ρωσία. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα της Ρωσίας πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά και ότι θα έπρεπε να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ εγώ να σας εξηγήσω γιατί το θέμα αυτό είναι τόσο σημαντικό από πολιτικής απόψεως και οικονομικής. Κοιτάξτε, εννοείται ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λαμβάνουν χώρα συζητήσεις στο Συμβούλιο, το θέμα των κυρώσεων και των επιπτώσεων. Είναι ένα θέμα που φυσικά βρίσκεται εν εξελίξη ακόμα. Επανέρχομαι λοιπόν στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στα περιβαλλοντικά αγαθά. Πρόκειται για θέμα που αφορά άμεσα την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομία και η Μόνικα μας, ε, Χένσκι θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε για να σας παρουσιάσω αυτή την πρωτοβουλία. Πολλοί ίσως από εσά το γνωρίζετε γιατί συζητήσαμε τα Green Goods και στο παρελθόν έγινε μια ακρόαση πέρυσι και έγιναν πολλές ανταλλαγές ε, απόψε με το Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Αλλά ε, να σας ενημερώσω για τις διαπραγματεύσεις της 8ης Ιουλίου που έλαβαν χώρα στη Γενέβη, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με 13 άλλα ε, κράτη, με 41 χώρες δηλαδή συνολικά, ε, έκαναν σημαντικά βήματα για την εμπορία πράσινων αγαθών και ε, τεχνολογιών. Ε, ο σκοπός είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι επωφελής όχι μόνο για το εμπόριο αλλά και για το περιβάλλον και για τις κλιματικές αλλαγές και θα ενθαρρύνει τις καινοτομίες καθώς επίσης θα δώσει απάντηση ε, σε θέματα νέων τεχνολογιών υπάρχει η μόνιμη δέσμευσή μας για την ε, ε, απελευθέρωση των, ε, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αλλά στο παρελθόν BA έχουμε μια ειδική αναφορά στην απελευθέρωση των πράσινων αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, στις διμερείς διαπραγματεύσεις μας προσπαθήσαμε πάρα πολύ να έχουμε μια εμπροστοβαρή προσέγγιση για την απελευθέρωση αυτών των αγαθών και υπηρεσιών, όπως παραδείγματος χάρη Σιγκαπούρη έχουμε συνάψει μια τέτοια συμφωνία. Εδώ θα έχουμε ε, μια πολυμερή συμφωνία με 40 συν μέλη του ΠΟΕ που όχι μόνο θα απελευθερώσει τα πράσινα αγαθά και υπηρεσίε αλλά θα ενισχύσει και το σύστημα του ΠΟΕ. Γιατί ακριβώ μιλάμε. Είναι ένα μάλλον τεχνικό θέμα. Έχω μια παρουσίαση που θα κυκλοφορήσει στα μέλη σα. Θα χρησιμοποιήσω κάποιε από αυτέ τι διαφάνειε αλλά μπορείτε να δείτε και τι περισσότερε λεπτομέρειε στην παρουσίαση, την ε, πλήρη όλα τα μέλη του ΠΟΕ χρειάζονται καλύτερη και φθηνότερη ε, πρόσβαση σε περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες και τεχνολογίες. Τι είναι αυτά. Είναι αυτά που χρειάζονται ή περιλαμβάνονται σε διαδικασίες που αφορούν την αντιμετώπιση της μόλυνσης του αέρα, ε, της ε, ε, επεξεργασίας αποβλήτων για την τεχνολογία πόσιμου νερού κλπ. κλπ. Είναι μια ευρύτατη γάμα προϊόντων που συμβάλλουν άμεσα στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, στο πρόβλημα στην επίλυση δηλαδή των προβλημάτων αυτών, στην αηφόρο ανάπτυξη κλπ. Ελπίζουμε να καταργήσουμε τα, τους δασμούς ε, για τα προϊόντα αυτά με την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων. Ιδανικά όμως δεν θα έπρεπε να σταματήσουμε σε αυτό το στάδιο. Στο μέλλον θα θέλαμε να έχουμε μια συμφωνία που θα καλύπτει και, τις και τα μη δασμολογικά εμπόδια και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Αν θέλουμε να Έχουμε πράσινη ενέργεια. Δεν χρειάζεται απλώς να αγοράσει κανείς μια αεροτουρμπίνα. Χρειάζεται να έχει πρόσβαση και στις παρέτητες υπηρεσίες, στις μηχανολογικές και συμβουλευτικές. Γι' αυτό η, η πρόθεση μας δεν είναι μόνο να απελευθερώσουμε τους δασμούς ε, για τα αγαθά, αλλά σε μεταγενέστερη φάση να περιλάβουμε και τις υπηρεσίες και διαπραγματεύσεις για μη δασμολογικούς φραγμούς. Μια εκτιμήση δείχνει ότι 65% αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες είναι, στις αγορές, συγγνώμη, είναι υπηρεσίες και 35% μόνο είναι αγαθά. Και οι περισσότεροι παρέχουν και αγαθά και υπηρεσίες από τους παρόχους. Αυτή η πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μας, θα έχει πολύ συγκεκριμένα ωφέλη και θα αναφέρω έξι από αυτά εδώ. Πρώτον, η πρωτοβουλία αυτή θα προωθήσει το παγκόσμιο εμπόριο πράσινων αγαθών και υπηρεσιών. Η αγορά αυτή ε, εκτιμάται ότι είναι ένα τρισεκατομμύριο αλλά υπάρχει, σύμφωνα, μα θα υπάρχει σύμφωνα στις μελέτες μια αγορά 2-3 εκατομμυρίων μέχρι το 2020. Ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές ε, υπάρχει ε, αύξηση της ζήτησης. Σίγουρα η πρωτοβουλία αυτή θα προωθήσει την, την πράσινη βιομηχανία παγκοσμίω, αλλά ιδίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε μια ε, εργατική δύναμη ε, και η πράσινη βιομηχανία βιομηχανία όχι μόνο θα δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά ιδίω σε μια περίοδο ανα... θα δημιουργηθούν περισσότερε θέσει εργασία σε αυτόν τον τομέα. 4 εκατομμύρια θέσει εργασία ε, αφορούν οι υπηρεσίε αυτέ και τα αγαθά σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, έχουμε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα ε, όπως ξέρετε, ε, υπάρχει μια πρόταση κομισιόν για ένα πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα και επίσης θα υπάρχει πρόσβαση σε φθηνότερες τεχνολογίες με σκοπό να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας που όλοι ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν στη νέα συμφωνία για το κλίμα και που θα διαπραγματευτούμε στο τέλος του 2015 στο Παρίσι. Τέταρτον, φθηνή πρόσβαση στις τεχνολογίες. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τους αναπτυσσόμενους εταίρους μας. Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει ήδη κάποιες αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι σημαντικό ότι η Κίνα από την αρχή είναι συμβαλόμενο μέρος. Αν δείτε τα 40 μέλη της πρωτοβουλίας αυτής, ε, ε, κάποιες από αυτές ε, ε, καλύπτουν, έχουν την κρίσιμη μάζα. Επίσης υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες όπως είναι η Κωνσταντίνα και ελπίζουμε ότι και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες θα συνειδητοποιήσουν τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει αυτή η συμφωνία και θα έρθουν στις διαπραγματεύσεις. Πέμπτον, και νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία, ε, αμέσως μετά τη συζήτηση για τη Ρωσία και την ανατολική ε, σχέση γειτονίας, θα διασφαλίσει η συμφωνία αυτή την, ε, τον εφοδιασμό με ενέργεια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μειώσει την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Την συμφωνία υποστηρίζουν όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Ομπάμα ε, συμπεριέλαβε τη συμφωνία αυτή στο δικό του σχέδιο για το κλίμα και η Κίνα, όπως σας είπα, ήδη συμμετέχει, ε, γιατί είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή για τους στρατηγικούς του στόχους και για την αντιμετώπιση της ρήπανσης της ατμόσφαιρας. Και εκτών είναι πολύ σημαντικό η νέα όθηση που θα δώσει η πρωτοβουλία αυτή στον ΠΟΕ. Νομίζω ότι είναι στην περίοδο μετά τον Πάλι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμό Εμπορίου να ε, τεθεί σε εφαρμογή η ε, εντολή που έχουμε για τα πράσινα αγαθά και υπηρεσίες και η πρωτοβουλία κάνει ακριβώς αυτό. Είναι ανοιχτή η πρωτοβουλία για όποια χώρα θα ήθελε να συμμετάσχει. Είναι σημαντικό ότι ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΕ καλωσόρισε την πρωτοβουλία αυτή όταν ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου. Τα επόμενα βήματα ποια είναι. Τα επόμενα βήματα ήδη αναφέρθηκαν από τον αξιότιμο κύριο Πρόεδρο Όσον αφορά τους γύρους διαπραγματεύσεων, θα έχουμε το δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι αρχική γύρη διαπραγματεύσεων. Συζητάμε την προσέγγιση ε, μέσω της οποίας θα προχωρήσουμε στις πραγματικές ε, διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, πιστεύουμε, στις αρχές της ερχόμενης χρονιάς. Η δημόσια διαβούλευση έκλεισε, θα δημοσιευτεί η σχετική έκθεση. Επίσης θα κάνουμε μια ε, μελέτη αντικτύπου και αηφορίας μέσα στα πλαίσια του SIA θα εξετάσουμε το οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών και ε, αυτός είναι ένας καλός υποψήφιος από την πλευρά την περιβαλλοντική. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, κοινωνία των πολιτών, η βιομηχανία ε, συμμετείχαν ε, στη Γενέβη και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον και περιμένουμε να ε, δούμε τη συζήτηση και τα, τις που θα έχει να θέσει στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας κάνετε για να ξέρουμε πώς ακριβώς έχει τοποθετηθεί το θέμα από μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά βεβαίω και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το ΕΛΚ έχει ερώτηση. Σοσιαλιστέ, Ούτε από εκεί βλέπω ερώτηση. Α, ο κύριος Κάσπα. Ευχαριστώ πολύ. Έλειπα από τη θέση μου. Ήθελα να σας πω ότι πραγματικά δεν ξέρω τι θέση να πάρω. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που με μεγάλη δυσκολία μπορεί καταρχήν να βρει ορισμό για το τι είναι προϊόν περιβαλλοντικό και τι δεν είναι, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από αυτή την κατηγορία. Θεωρώ πραγματικά ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους δασμούς για όλα τα προϊόντα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για οτιδήποτε δεν πλήττει το περιβάλλον και προωθεί τις εμπορικές συναλλαγές και την οικονομική μας σχέση. Βεβαίως, αν δούμε ότι άλλες περιοχές του κόσμου οικειοθελώς έχουν μειώσει αυτούς τους δασμούς και έχουν υιοθετήσει τέτοια ευνοϊκά μέτρα, τουλάχιστον θα μπορέσουμε κι εμείς ή θα έπρεπε να μπορέσουμε να θέσουμε σαν στόχο την αμοιβαιότητα. Κάποιος από τους ε, σοσιαλιστές θέλει να κάνει ερώτηση. Όχι, στην συντηρητική. Άλντε, πιλελεύθερη. Γκουέ. Ο Μπέντ. Είναι σωστό αυτό που είπε ο Ντάνιελ ε, Κάσπαρη. Δεν είναι εύκολο κανείς να θεωρήσει ποιο είναι και ποιο δεν είναι προϊόν που μπορεί να μπει στην κατηγορία των ε, περιβαλλοντικών αγαθών. Οι εκτιμήσεις, αν θέλετε, είναι ένα θέμα όσον αφορά το περιβαλλοντικό χαρακτήρα αυτό των προϊόντων. Απ' την άλλη πρέπει να δούμε και το οικονομικό κομμάτι και αν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε τι έκαναν κάποια άλλα κράτη, κάποιες άλλες περιοχές και στα πλαίσια του ΠΟΕ αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δει εάν γενικότερα στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές δεν θα πρέπει να μπει μια περιβαλλοντική συνιστόσα έτσι ώστε οι ροές και οι ανταλλαγές των προϊόντων να οργανωθούν με έναν τρόπο. Βλέπουμε πολλές φορές ε, κατηγορίες προϊόντων που βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτή την κατηγορία των ε, περιβαλλοντικών αγαθών. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα, να δώσουμε όθηση σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια πιο σωστή, πιο ισορροπημένη πολυμερή συμφωνία. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, μια δεύτερη παρατήρηση. Αναφερθήκατε στον τομέα των υπηρεσιών, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν σημαντικό τομέα αυτής της συμφωνίας. Βεβαίως υπάρχουν όμως εδώ πολύ συγκεκριμένες ε, ευαίσθητες ε, περιοχές παραδείγματος χάρη το νερό η παροχή ύδατος ξέρετε παραδείγματος χάρη το καθεστώς που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει κάτι παρόμοιο εδώ στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται να το δεχθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δηλαδή να υπάρχει ιδιωτική διαχείριση και διευθέτηση στον τομέα του νερού, παραδείγματος χάρη. Αυτό όμω βέβαια είναι μια άλλη συζήτηση. Ο Γιάννικ. Ευχαριστώ. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Είναι πάντοτε ενδιαφέρον να υπενθυμίζουμε ότι είναι ένας τομέας ε, δεν έχει πληγεί τόσο πολύ από την κρίση, αλλά δημιουργεί ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας παρόλα τα όσα λέγονται στα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό που είναι δύσκολο σε αυτή την πρωτοβουλία είναι να κρίνουμε, να σταθμίσουμε την αξιοπιστία της και την ειλικρίνειά της θα έλεγα. Βλέπουμε πολύ καλά ότι αν ο στόχος είναι πραγματικές πράσινες τεχνολογίες που επιτρέπουν την καταπολέμηση κατά της ε, κλιματικής αλλογής, στην, στην ομόνωση των κτηρίων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε πρέπει να είμαστε υπέρ, να, είμα, να είμαστε ευνοϊκοί όχι μόνο για αυτή τη συμφωνία, αλλά αν ταυτόχρονα μπορούμε στα φωτοβολταϊκά να καταπολεμήσουμε το dumping το Κινέζι, των Κινέζων, πράγμα που δεν κατόρθωσε η Ευρώπη. Ενώ έχουμε απόδειξη ότι οι παραγωγοί ε, Κινέζοι παρακάμπτουν το ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, και αν μπορούμε επίσης να καταπολεμήσουμε την επιδότηση των ορυκτών καυσίμων. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε βάζουν το θέμα αυτό στο τραπέζι, τις διαπραγματεύσεις και εμείς ε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και υπάρχει το θέμα των καταλόγων. Ένας αντιδραστήρας πυρηνικός είναι περιβαλλοντικό αγαθό, προϊόν. Λέτε ναι. Εγώ λέω όχι. Ένας, ε, ε, ένα, για την καύση των, των αποβλήτων, ίσως η, ε, το έλαιο κοκοφίνικα είναι περιβαλλοντικό αγαθό. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές εκτιμήσεις, αλλά ο στόχος είναι να ευνοήσουμε τεχνολογίες ε, που ε, θα θέλουμε να κάνουμε τους άλλους να πιστέψουν ότι είναι πράσινες ενώ δεν είναι. Είναι θέμα τέχνασμα επικοινωνίας και σε όλες ε, τις διαπραγματεύσεις των ΠΟΕΝ υπάρχει ένα άλλο θέμα, είναι το θέμα των ε, των επεξεργασιών ε, στην παραγωγή. Αν πάρουμε τον έλαιο του κοκοφίνικα, αν πάρουμε το τελικό προϊόν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ρηπαίνει λιγότερο από το γκαζόιλ, από την βενζίνη. Αν πάρετε όλη την διαδικασία παραγωγής, δεν είναι περιβαλλοντικό αγαθό. Και αυτή είναι η συζήτηση που είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση ε, με τα αγροκαύσιμα. Μπορεί να είναι μια πρωτοβουλία ενδιαφέρουσα αν είμαστε σοβαροί ως προς τον κατάλογο. Και δεύτερον, αναφέρατε τις αναπτυσσόμενες χώρες και έχετε δίκιο ως προς την κλιματική αλλαγή. Το θέμα είναι ότι συνολικά, γενικά, οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι σε αυτήν την πρωτοβουλία. Σε αυτήν την πολυμερή ε, πρωτοβουλία θα επιβάλλουμε, αν είναι καλή η συμφωνία, θα επιβάλλουμε την ρήτρα της, ε, ε, της πιο ευνοημένης χώρας ούτως ώστε οι χώρες να μπορούν να προσχωρήσουν σε αυτά τα περιβαλλοντικά αγαθά. Η ιδέα στο κείμενο είναι καλή ιδέα, η βασική ιδέα, αλλά θα γίνει αξιόπιστη μόνο αν είμαστε σοβαροί για το περιβάλλον και αν δεν είναι ένας άλλος τρόπος να πουλήσουμε προϊόντα και ε, υπηρεσίες που παρόλη την επικοινωνία είναι αντίπαλοι, είναι εχθροί της προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Συμμεριζόμαστε την προβληματική σχετικά με τον κατάλογο των εμπορευμάτων που θέλουμε να περιληφθεί ε, στη λίστα αυτή για λόγους που μόλις αναφέρθηκαν. Επίσης προσθέτουμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και επικίνδυνο, γιατί θα μπορούσαμε να κατακλειστούμε από προϊόντα που θα προέρχονται από την Κίνα και από την Νοτιοανατολική Ασία σε τιμές ε, πολύ ανταγωνιστικές, που δεν θα σέβονται όμως τους κανόνες ασφάλειας, αλλά και κατασκευής. Ε, δεν θέλουμε να διευκολύνουμε έτσι ε, τις χώρες αυτές που θέλουν να υποφεληθούν από την αγορά εργασίας, τις διαφορές στην αγορά εργασίας, ε, με αθέμητο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε και κυρίως από ποιον παράγεται και πώς. Ευχαριστώ. Κανένα άλλο δεν ζητάει το λόγο. Μπορείτε να απαντήσετε. Θα αρχίσω λέγοντας ότι είμαι από τη Βουλγαρία. Για μένα ε, το καταφατικό νεύμα του κεφαλού είναι το αντίθετο από το δικό σας λοιπόν. Ε, βάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις σας για τις οποίες σας ευχαριστώ. Καταρχάς να ξεκινήσουμε τα προϊόντα. Τι είναι ε, περιβαλλοντικό προϊόν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις τεχνικές προκλήσεις που αναφέρατε. Δεν θα είναι εύκολο. Ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε πολύ ρεαλιστές ε, στις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε μεγάλες ακαδημαϊκές συζητήσεις γιατί τέτοιες προσπάθειες απέτυχαν στο παρελθόν στον ΠΟΕ. Υπάρχει μια επιτροπή στον ΠΟΕ που διαπραγματεύτηκε και συζητούσε επί χρόνια τα θέματα αυτά και δεν οδήγησε η συζήτηση αυτή σε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την απελευθέρωση του εμπορίου. Βέβαια, την άλλη μεριά, κανεί δεν, θα μπορεί, δεν θα μπορεί να προτείνει ένα προϊόν χωρί ε, να το υποστηρίζει με βάσιμη ε, επιστημονική και τεχνική επιχειρηματολογία και οι άλλοι θα, μπορούσαν, θα μπορούν να αντιταχθούν. Ε, και για κάθε συζήτηση θα υπάρχουν εμπειρογνώμονες από τα Ηνωμένα Έθνη, από το πρόγραμμα για το περιβάλλον, από περιβαλλοντικές NGOs, από think tank κλπ. Ε, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα καταλήξουμε με ένα κατάλογο που θα έχει όχι μόνο οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά ωφέλη. Τώρα για το θέμα των υπηρεσιών. Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα σε δύο είδη υπηρεσιών. Τις παραδοσιακές περιβαλλοντικές υπηρεσίες, πούμε για τη διαχείριση των υδάτων. Κάποιες από αυτές ε, τις ε, υπηρεσίε κάποιε από αυτές συζητούνται στι διαπραγματεύσει ΤΙΣΑ για τι υπηρεσίε. Αλλά αυτό θα, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ. Είναι υπηρεσίε που σχετίζονται άμεσα με κάποια αγαθά. Παραδείγματο χάρη εγκατάσταση, ε, συντήρηση, μηχανολογική υποστήριξη κάποιου περιβαλλοντικού προϊόντο. Εδώ υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά θεωρούμε ότι με τι τεχνικέ συζητήσει ίσω στο μέλλον σε μια μελλοντική φάση, θα έχουμε και ε, την απελευθέρωση αυτών των επικουρικών ε, υπηρεσιών όπως τις λέμε. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ανέφερα κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και έχουμε ενδιαφέρον ε, και από άλλες χώρες. Είχαμε συζητήσει με κάποιους εταίρους μας στη, στη Βόρεια Αφρική, το Μαρόκο παραδείγματος χάρη. Είχαμε κάποια εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Χίλη κάναμε συζητήσεις με το Μεξικό. Ε, κάνουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια να φέρουμε, να προσελκύσουμε ε, όσο γίνονται περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, αλλά ε, ό,τι γίνει θα γίνει ε, πίεση όσον αφορά ε, τη δασμολογική κλίμακα και η συμφωνία θα είναι ανοιχτή ε, για όποιον θέλει να συμμετάσχει στο μέλλον. Από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών ε, αυτό μπορεί να έχει ενδιαφέρον και από την άποψη των εξαγωγών και από την άποψη των εισαγωγών. Ε, ο εκπρόσωπος της Κώστα Ρίκα, παραδείγματος χάρη, είπε ότι όταν συμμετέχει άρχισε να συμμετάσχει στην σχετική συμφωνία η Κωνσταντίνα ε, για τις ε, τεχνολογίες της πληροφορικής. Δεν ε, είχε καθόλου τέτοια παραγωγή, αλλά έκτοτε άρχισε να παράγει και έγινε εξαγωγέας υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής. Τώρα, γιατί γίνονται οι διαπραγματεύσεις αυτές στον ΠΟΕ. Είναι και αν θα είναι διμερής ή πολυμερής η συμφωνία. Ελπίζουμε πάρα πολύ ότι θα γίνει πολυμερής. Όπως ανέφερα όμως, ε, το plurilateral θα ενισχύσει το multilateral, ε, γιατί ε, οτιδήποτε αποφασιστεί, εφόσον θα είναι στα πλαίσια του ΠΟΕ, θα είναι δεσμευτικό όσον αφορά τους δασμούς. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν θα είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, ε, δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Ας πούμε δεν θα λύσουμε το πρόβλημα των βιοκαυσίμων, δεν θα λύσουμε το όλο πρόβλημα των μεθόδων παραγωγής. Αλλά αν ξαναεστιάσουμε πιστεύω σε ένα υποσύνολο προϊόντων, η χρήση των οποίων μπορεί να συμβάλλει σε διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν στην βελτίωση του, της προστασίας του περιβάλλοντος ή στην αντιμετώπιση των ε, κλιματικών αλλαγών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε κάποιους αναπτυσσόμενους εταίρους μας, αυτό θα είναι ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε και φυσικά με μεγάλη προσοχή θα παρακολουθήσουμε όλες ε, τις ε, ενεξελίξεις και συνεχιζόμενες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις. Φυσικά όλα αυτά που ακούσατε σήμερα θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, και στις περαιτέρω ε, συνομιλίες σας, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να σας ξαναδούμε και να συνομιλήσουμε μαζί σας. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και με το σημείο 15 και περνάμε στο 16. Το θέμα αυτό αφορά τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Acting Deputy Director General ο οποίος είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο οποίος βέβαια έχει και πολλές άλλες αρμοδιότητες αλλά έχει και την αρμοδιότητα του επικεφαλής ε, ήταν μάλλον ήταν ε, επικεφαλής των διαπραγματεύσεως του ΣΥΤΑ Λέω ήταν γιατί φυσικά έχει ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και θα κυρωθεί από ό,τι ξέρω στις 25 Σεπτεμβρίου. Αρχικά είχε δοθεί το πράσινο φως σε πολιτικό επίπεδο πέρσι τον Οκτώβριο. Προετοιμάστηκε ένα κείμενο, πιστεύω με μεγάλη επιτυχία, συγχαρητήρια λοιπόν. Και είμαστε πραγματικά πολύ περίεργη να δούμε όλα τα στοιχεία που καταφέρατε να συμπεριλάβετε σε αυτό το κείμενο. Ξέρω ότι υπήρχαν πάρα πολλά επίμαχα σημεία. Δώστε μας λοιπόν κάποιες πληροφορίες και για το περιεχόμενο της συμφωνίας και κατόπιν θα ακολουθήσουν συζήτηση για την ε, εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και σας δίνω το λόγο. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που επανέρχομαι στην Επιτροπή, στην τελευταία της ε, μετενσάρκωση. Πολύ ευχαρίστω να σας ενημερίσω πού βρισκόμαστε για την ΣΥΤΑ. Να σας πω σε... όσον αφορά την Συμφωνία ΣΟΕΣ δηλαδή, να σας πω ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα. Και επί τη ουσία τώρα θα ε, με καθοδηγήσετε εσείς για το ποια σημεία θέλετε να συζητήσουμε πιο λεπτομερώς, ε, κοιτάζοντας και την ώρα. Ε, πρόεδρε, ήδη αναφερθήκατε σε κανένα δύο θέματα για τα οποία ενδιαφέρονται τα μέλη της Επιτροπής σας. Σας πω ότι τελειώσαμε τις διαπραγματεύσεις τέλος Ιουλίου, στις 31 Ιουλίου ακριβώς. Έχουμε ένα πλήρες κείμενο αυτή τη στιγμή που έχει αποσταλεί στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για να το ε, εξετάσουν. Ο Καναδάς έστειλε το κείμενο στις επαρχίες του θα κάνουμε μια συζήτηση αυτού του κειμένου με τα κράτη-μέλη στις 12 ε, Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή ε, εμπορικής πολιτικής σε επίπεδο τακτικών μελών. Ο στόχος είναι ο κύριος Μπαρόζο και ο Πρωθυπουργό του Καναδά να ανακοινώσουν επίσημα την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στις 26 Σεπτεμβρίου στην Οτάβα, στο Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Μετά θα περάσει από, νομική, ε, από νομικό χτένισμα ε, το κείμενο αυτό και από τη διαδικασία των μεταφράσεων θα χρειαστεί να είναι ε, αυθεντικό το κείμενο σε όλες τις ε, ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο Καναδάς φυσικά για λόγους ε, συνταγματικού θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο γαλλικό κείμενο. Είναι ένα σύνθετο κείμενο, καινοτόμο από πολλές ε, απόψεις, άρα οι νομικοί θα έχουν περισσότερο να πούν από ό,τι κάνουν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις και θα είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα το υποβάλουμε το κείμενο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για έγκριση. Για την ουσία τώρα, να υπενθυμίσω εν συντομία κάτι το οποίο ήταν κοινό τόπο στι διαπραγματεύσει όταν ξεκινήσαμε. ήταν κοινό τόπο, αλλά εντωμεταξύ ε, ξεχάστηκε κάπω. Η συμπληρωματικότητα δηλαδή των οικονομιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Καναδά. Ε, ο Καναδάς έχει μια οικονομία που μοιάζει εντυπωσιακά με κάποιες οικονομίες των κρατών μελών. Ε, ισχυρός εμπορικός εταίρος, εξαγωγέας, επενδυτής. Ε, το διεθνές εμπόριο έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την ευημερία του Καναδά, πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλες χώρες με μεγαλύτερη εσωτερική αγορά. Επίσης, ο Καναδάς είναι μια, ένας ιδιαίτερα ισχυρός επενδυτής στην Ευρώπη. Η οικονομία του Καναδά είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συγκρίση με κάποια κράτη-μέλη η οικονομία ε, του Καναδά, αλλά ο Καναδάς ε, επενδύει στην Ευρώπη πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές του κόσμου και επενδύει ε, πάνω από τα διπλάσια από ό,τι επενδύουμε εμείς στην, στον Καναδά. Οι Καναδοί ε, λοιπόν επενδυτές ε, είναι αναπόσπαστο μέρος του οικονομικού συστού. Δημιουργούν ε, ευημερία, δημιουργούν απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτό σας δίνει μια ιδέα για το πόσο σημαντικός είναι ο Καναδάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικός και αναπόσπαστος είναι ο Καναδάς για την οικονομία της Βόρειας Αμερικής. Ταυτόχρονα όμως ε, η Ανατολική Ασία παρέχει κάποια εναλλακτική ε, λύση, αλλά κάπως άβολη, όπως ξέρουμε και εμείς από τις σχέσεις μας με την Ανατολική Ασία. Ο φυσικός εταίρος του Καναδά είναι η Ευρώπη. ο Καναδάς εισάγει όχι τόσο πρώτες ύλες, γιατί είναι πλούσιος ε, σε πρώτε ύλε, αλλά ενδιάμεσα προϊόντα, υπηρεσίε, μηχανολογικό εξοπλισμό, για να μην αναφέρω και καταναλωτικά προϊόντα, όλα αυτά είναι υπέρ τη ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Οικονομία. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμπληρωματικότητα λοιπόν και σε όλε αυτέ τις διαπραγματεύσει κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε μαζί με ε, τους καναδού συνομιλητέ μα για να ενισχύσουμε αυτή τη συμπληρωματικότητα στην ανταλλαγή παραχωρήσεων. Για τα αγαθά και και τους δασμούς. Η συμφωνία αυτή θα απελευθερώσει τους δασμούς ε, στο 99% σχεδόν για ε, όλα τα αγαθά. Ε, απελευθέρωση το πολύ μέσα σε 7 χρόνια. Παρ' όλα αυτά και οι δύο πλευρές έχουν διατηρήσει την προστασία για καμιά δεκαριά πολύ ευαίσθητα προϊόντα. Λίγα ευαίσθητα προϊόντα στο γεωρικό τομέα. Ε, διανοητική ιδιοκτησία, κατά παράδοση, κριτικάρεται ο Καναδά ότι έχει χαμηλότερα στάνταρα από ό,τι άλλε αναπτυγμένε χώρε. Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει μια αμοιβαία ικανοποιητική ε, συμφωνία, καλύτερη προστασία του copyright, καλύτερη ε, εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία, καλύτερη προστασία για τα φαρμακευτικά προϊόντα και για τι γεωγραφικέ ενδείξει ε, ανοίξαμε καινούργιε προοπτικέ. Όσον αφορά τι υπηρεσίε και τι τις επενδύσεις και την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Πάλι ε, είναι καινοτόμα η συμφωνία αυτή. Είναι DDA+, δηλαδή ενώ και εμείς και ο Καναδάς είμαστε από τα φιλόδοξα μέλη του ΠΟΕ, ανακοινώσαμε ότι είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε στο DDA και τα δύο μέρη έχουν παρόμοιες ευαισθησίες και παρόμοιου τομείς που θέλουν να προστατεύσουν ε, δημόσιες υπηρεσίες, η ΔΕΚΟ ε, στη δική μας ορολογία, όπου διατηρήσαμε το ίδιο, ε, τον ίδιο βαθμό ευελιξίας όπως και με τους πολυμερείς κανόνες. Ο πολιτισμός είναι ένα άλλο θέμα. Ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον πολιτισμό δεν είναι ακριβώς ο ίδιο στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ήταν αρκετά πολύπλοκο θέμα αλλά συμφωνήσαμε σχεδόν αμέσως επί της ουσίας στο τι θέλαμε να επιτύχουμε. Κρατήσαμε την παραδοσιακή μας ε, προσέγγιση για τα οπτικοακουστικά. Διατηρήσαμε κάποια πλεονεκτήματα, παραδείγματο χάρη είναι καλύτερη προστασία του copyright για τους ε, πολιστικούς operators. Έχουμε καλύτερη μεταχείριση στον Καναδά όσον αφορά τον έλεγχο των επενδύσεων από ότι επενδυτέ από άλλε χώρε, λαμβάνοντα υπόψη ότι στην Ευρώπη δεν ελέγχουμε τι επενδύσει παρά μόνο για λόγου εθνική ασφάλεια. Η προστασία των επενδύσεων. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι όπως ξέρουμε αυτό είναι ένα από τα πιο αφιλεγόμενα κομμάτια που δημιούργησαν τις περισσότερες συζητήσεις και σίγουρα θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ε, ε, είμαστε στο τελευταίο ε, στάδιο των εξελίξεων. Ξεκινήσαμε από το κεκτημένο σε κράτη, στα κράτη-μέλη. Ξεκινήσαμε από τη στιγμή που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υιοθέτησαν ε, τον μεταβατικό κανονισμό για τις επενδύσεις μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Λάβαμε υπόψη μας τις εξελίξεις της δημόσιας συζήτησης μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα αυτό που επιτύχαμε που απαντάει σε πολλές από αυτές τις ανησυχίες. Είναι η τελευταία λέξη. Δεν, δεν είναι ε, βέβαια... Ε, δεν έχει μπει ακόμα η τελευταία λέξη. Μέχρι εδώ έχουμε φτάσει, αλλά η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Ε, είχαμε πάντως την σχετική διαπραγματευτική εντολή ήδη πριν από μερικά χρόνια. Για τις ε, ε, προμήθειες του δημοσίου. Ε, διασχίσαμε νέα σύνορα με τη συμφωνία αυτή στον τομέα αυτό. Κάποιες από τις λίγες ε, αγορές που δεν ήταν ανοιχτέ στο δημόσιο στο διεθνές εμπόριο έχουμε γι' αυτό καταπληκτικά αποτελέσματα. Προσφέρουμε στον Καναδά πρόσβαση στις εσωτερικές μας προμήθειες του δημοσίου. Ανταποκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο ο Καναδάς. Ε, η αμοιβαιότητα δεν είναι η ίδια ακριβώς με αυτή που προσφέρουν μεταξύ τους τα κράτη-μέλη, αλλά είναι αρκετά κοντά σε αυτό. Είναι πολύ ισορροπημένη η ανταλλαγή ε, παραχωρήσεων. Οι κανόνες είναι GPA+, και εμείς και ο Καναδάς ε, θέλουμε πάρα πολύ οι κανόνες για τις προμήθειες του δημοσίου να είναι διαφανείς, δίκαιοι και εύχριστοι από τις δημόσιες αρχές και από τις δύο πλευρές και νομίζω ότι έχουμε βασιστεί στους ε, ε, πολυμερείς κανόνες που υπήρχαν από αυτού. Ε, η συμφωνία αυτή λοιπόν είναι συγκρίσιμη με το GPA Plus και δίνει πρόσβαση στις αγορές του δημοσίου πολύ παραπάνω από ό,τι ισχύει στο παρελθόν. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν εκτεταμένες διατάξεις ε, για μη διασμολογικά μέτρα, ε, για την κανονιστική συνεργασία. Έχουμε κανόνες που θα ενισχύσουν την διαφάνεια, που προωθούν την εσωτερική νομοθεσία. Δρεώνουμε την καλή συνεργασία που είχαμε με τον ε, Καναδά σχετικά με υγειονομικά θέματα. Θα έχουμε ε, μια αναγνώριση ε, προτύπων και υποσχέσεις ε, περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον. Καλό επίσης κεφάλαιο για την αηφόρο ανάπτυξη όπου υπήρχε άμεση συμφωνία για την ουσία και μετά μακρές διαπραγματεύσεις για το πώς να συμφιλιώσουμε τις διάφορες προσεγγίσεις περίπλοκες ε, βεβαίως αυτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά νομίζουμε ότι ήταν επιτυχημένες και ο τρόπος ε, με τον οποίο συμβιβάσαμε τις διάφορες προτάσεις θα βελτιώσει την λειτουργία αυτής της συμφωνίας ε, και μας έδωσε πάρα πολλές χρήσιμες ιδέες για άλλες διαπραγματεύσεις με άλλους εταίρους, κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτές, αυτά είναι τα πλεονεκτήματα Επίσης στείλαμε στο Κοινοβούλιο την ίδια αξιολόγηση που στείλαμε και στα κράτη-μέλη. Δεν είναι πλήρη. Στον Αύγουστο ακόμα στα προσπαθούσαμε να οριστικοποιήσουμε τα νομικά κείμενα για να μην υπάρχουν λάθη στα κείμενα και νομίζω ότι πάρα πολλοί θα ανακαλύψουν ότι αφήσαμε ακόμα πάρα πολύ λάθη στο κείμενο. Ε, δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο για περισσότερη οικονομική ανάλυση, θα το πράξουμε όπως ξέρουμε όλοι, ε, το κείμενο έχει διαρρεύσει, είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, είναι λυπηρό. Ε, βεβαίως θα δημοσιεύσουμε εμείς το κείμενο αυτό, θέλαμε απλώς να έχουμε λίγο χρόνο ούτως ώστε όσο το δυνατόν περισσότερο να διορθώσουμε τα λάθη και έπρεπε να μιλήσουμε με τους Καναδούς φίλους μας ε, διότι δεν είναι κάτι που πρέπει κανείς να το δημοσιεύσει μονομερός χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου. Θα το συζητήσουμε λοιπόν με τον Καναδά και θα δημοσιεύσουμε το κείμενο. Ε, βεβαίως ε, το, η εργασία συνεχίζεται δεν χρειάζεται αναθεώρηση νομική, αλλά είναι σημαντικό όλοι να μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση σε ένα κείμενο που έχει λάβει και τη συγκατάθεση του Καναδά. Βεβαίως εσείς και τα μέλη θα με καθοδηγήσετε για οποιαδήποτε βελτίωση ε, θέλετε να επιφέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζητήσω πρώτα από τις ομάδες. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα μας δίνετε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψη για το θέμα αυτό. Είναι εντυπωσιακή η εργασία που έχει κάνει η Επιτροπή όσον αφορά την συμφωνία αυτή με τον Καναδά. Αν οι πληροφορίες ευσταθούν, αυτές που σήμερα μας δόθηκαν, θεωρώ ότι όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες, όσον αφορά τα πρότυπα, όσον αφορά τα μειονικά θέματα, έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Εμείς έχουμε ζητήσει κάποια πράγματα, ελπίζω να έχουν συμπεριληφθεί. Εάν ναι, εάν συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο, στο έγγραφο, τότε βεβαίως ε, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί και να μην γίνει το ίδιο που έγινε και με την συμφωνία για τις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου υπήρχαν ε, σημαντικές αποκλήσεις μεταξύ των προτύπων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών που προέβλεπε η συμφωνία. Ελπίζω δηλαδή να μην γίνει κάτι όπως αυτό που έγινε με το κρέας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν σύμφωνα σημεία τα οποία έχουμε επισημάνει και τα οποία ελπίζουμε να έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία. Από την άλλη, Υπάρχει το θέμα της προστασίας των επενδύσεων, το έθιξε η Επιτροπή αυτό. Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις, κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες δίνουν εντολή για το θέμα της προστασίας των επενδύσεων. Ξέρουμε τη στάση του Καναδά. Με μεγάλη πλειοψηφία όμως, όταν εκφραζόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη από το 2010-2011, όταν άρχισε να ισχύει η Συμφωνία της Λισαβόνας, και στην έκθεση Καντέρ Αρίφ λέμε ότι σε περιπτώσεις διαμαχών που αφορούν τέτοιες επενδύσεις ζητούμε την παρέμβαση της ε, Επιτροπής και λέμε ότι εδώ δεν μας δημιουργεί πρόβλημα αυτή η προστασία των επενδυτών. Θέλω να πω ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές με το Συμβούλιο έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες και θα ήθελα ε, άσχετα με το αν είμαστε υπέρ ή κατά της προστασίας των επενδύσεων, να συμπληρωθεί εδώ αυτή η συμφωνία με αυτό τον τρόπο. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι σαφής. Έχουμε συμφωνήσει ομόφωνα για το θέμα της προστασίας των επενδύσεων και σας διαβάζω εδώ την έκθεση Καντέρ Αρίφ, αν δεν τη θυμάστε, η οποία πέρασε ομόφωνα από την Ολομέλεια επιπλέον από τις διαμάχες ε, τις διακρατικές θα πρέπει να υπάρχει εδώ επανάβαση της Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προστασία των επενδύσεων. Ξέρω ότι κάποιες πολιτικές ομάδες χαμογελούν διότι πάντα ήταν κατά κάποιες πολιτικές ομάδες έχουν εκφραστεί κατά. Όμως, επαναλαμβάνω, εγώ με δυσκολία θα δεχτώ ότι εδώ αυτή η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρακαμφθεί και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οποίας η θέση ε, δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει, αλλά από την οποία έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να προχωρήσει σε μια εργασία για το θέμα αυτό της προστασίας των επενδυτών δεν εκφράζει εδώ την άποψή της. Θέλω να ξέρω ποια είναι η στάση για τη συμφωνία με τον Καναδά, ποια είναι η συγκεκριμένη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω επίσης να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας παραδώσει εδώ κάτι το οποίο της έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Οι σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Δεν ε, θα το ανέφερα το θέμα. Έχει καλυφθεί ο Ντάνιελ. Με προκάλεσε όμως και πρέπει να πω ότι ε, θα, ε, αν εξετάστε τις πρόσφατα καναδικά ψηφίσματα που ψηφίστηκαν για την συμφωνία, είπαμε για τις διαφορές ότι ε, δεν ξέρω, σε μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο όρημα νομικά συστήματα, είπα ότι δεν θέλουμε ISDS. Βεβαίως αυτό ήρθε μετά την έκθεση Καντήρα ε, το, του Κοινοβουλίου. Σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι που η Επιτροπή εκτιμά και έχω κάποιες ανησυχίες, αλλά είναι ένα θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα. Είναι μεγάλος παραγωγός γενοσύμων ο Καναδάς. Βεβαίως ίσως ε, δεν ε, ε, μπορεί να μην είναι αληθινά αυτά τα οποία λέγονται στο διαδίκτυο, δεν σταματάει αυτό να χρησιμοποιούν διαδικασίες αδειοδότησης και οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής. Δεν ξέρω πώς όλα αυτά τα πράγματα θα και ε, δεν θα μπορεί να σταματήσει τίποτα τον Καναδά ε, να ε, στείλει. Επίσης για την αηφόρα ανάπτυξη είπατε η Κομισιόν ότι ε, σας αρέσει το, το κείμενο αυτό, χρειάζεται περισσότερη οικονομική ανάλυση, αλλά νομίζω ότι στον Συμφωνία για την Εργασία βλέπουμε την προσέγγιση με την ναύτα. Δεν ξέρω εμείς για την Συμφωνία Ναύτα υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, στο δικαίωμα το, το, το κεφάλαιο πρέπει να υπάρχει εποπτεία, πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση. Δεν ξέρω ε, αν είναι ανοιχτό ε, το θέμα όταν επισκεφθήκαμε ως αντιπροσωπεία τον Καναδά συζητήσαμε ε, με τις τοπικές κυβερνήσεις σχετικά με τις διευθετήσεις τις τοπικές, τις επαρχιακές ε, και αν υπάρχει μονοπόλιο, αν υπάρχει τρόπος αντικατά του ανταγωνισμού και δεν ξέρω αν αυτά όλα θα μπορούσαν να περιληφθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σχετικά με την πρόοδο αυτής της συμφωνίας που είναι πάρα πολύ φιλόδοξη ε, και που έχει πλεονεκτήματα όσο προς τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις, το ερώτημα που θα θέσω νομίζω ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση ε, στην υπογραφή. Προχώρησαν αρκετά στις διαπραγματεύσεις, αλλά μετά υπήρξε ένα κενό και κάποια καθυστέρηση. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι, μπορούμε να μάθουμε τίποτα εάν η ίδια η ναύτα θα πρέπει να τροποποιηθεί ε, σε σχέση με αυτήν την συμφωνία ή αν όλα είναι εγκεκριμένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, ε, τι συνεπάγεται για την ναύτα και ποιες είναι οι συνέπειες από την ναύτα και τι ε, σημαίνει για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κυρίως για ιατρικά προϊόντα. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Πολλά ακούστηκαν, αλλά θεωρώ ότι θα ανακαλύψουμε πολλά όταν δούμε το κείμενο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό εδώ να στείλουμε κάποια σωστά μηνύματα. Πολλοί παρακολουθούν αυτές τις διαπραγματεύσεις και περιμένουν πολλά για να δουν πώς εξελίσσονται οι διατλαντικές εμπορικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις και πιστεύω ότι θα ανοίξει ένας νέος ορίζοντας με επιπτώσεις που ίσως ακόμα δεν έχουμε φανταστεί. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ακριβώς επειδή πολλοί παρακολουθούν αυτήν την ε, συμφωνία οικονομικής και εταιρικής σχέσης τι δυσκολίες και διαφορές μπορούν να προκύψουν όπως παραδείγματος χάρη για το ISDS τις διαφορές και διαμάχες που μπορεί να προκύψουν. Το θέμα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Εδώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και εγώ ίδια θεωρώ ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί το καθεστώς που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα και να διασφαλίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλουμε με δυσανάλογο τρόπο αυτές ε, τις ε, διατάξεις, ιδίως για χώρες που δεν έχουν παρόμοιο καθεστώς. Και μια τελευταία ερώτηση. Οι μελλοντικές ε, ρυθμιστικές αποφάσεις πώς θα αντιμετωπιστούν από εδώ και πέρα από τις αρχές των δύο περιοχών, τις ευρωπαϊκές και τις καναδικές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω πολλές ερωτήσεις για διάφορα θέματα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ενημερωθήκαμε για την συμφωνία αυτή στις 6 Αυγούστου, την πρώτη εβδομάδα των διακοπών. Αμέσως προσπάθησα να, να καλύψω περισσότερα για την συμφωνία αυτή, αλλά όλοι είχαν πάει διακοπές και δεν υπήρχε κανείς να απαντήσει στις ερωτήσεις μου. Ε, επιπλέον, ο, ο μεγάλος αυτός αριθμός των ε, χιλιάδων απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση ε, είχαν δημοσιευτεί πριν ε, από δύο μόλις εβδομάδες. Ίσως τα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων αυτών έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στη Συμφωνία ΣΥΤΑ. Επιπλέον, το παρατηρητήριο ανακάλυψε ότι από τις 560 συναντήσεις με λόμπι οι 520, 92% δηλαδή, ήταν λομπίστες και μόνο 4% ήταν ομάδες που εξέφραζαν δημόσια συμφέροντα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Κομισιόν δεν ε, δίνει δεκάρα για τα δημόσια συμφέροντα, για τη δημόσια σφαίρα, παρά μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις χρηματοοικονομικές αγορές. Η ερώτησή μου είναι τι θα κάνετε για να πείσετε το Κοινοβούλιο ότι μπορεί να, να, ψηφίσει ε, την ε, συμφωνία αυτή όταν ε, ε, μεροληπτεί τόσο πολύ η Κομισιόν σχετικά με αυτούς που εκπροσωπεί. Πότε θα γίνει η δημόσια διαβούλευση για την ΣΥΤΑ και για την ΤΙΣΑ επίσης, είναι η άλλη ερώτηση. Ο Επίτροπος Δεχούχτ είπε πολύ συχνά ότι η συμφωνία αυτή είναι μια μεικτή συμφωνία και ότι θα υποβληθεί στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί δημιουργούμε ουσιαστικά μια κοινή αγορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό έχει νόημα. Ε, άρα, ε, η ερώτηση μου είναι η ΣΥΤΑ θα είναι και αυτή ε, ε μεικτή συμφωνία. Για το ISDS, την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους, μπορούν οι επιχειρήσεις στα δικαστήρια να ζητήσουν μεγάλες αποζημιώσεις για αποφάσεις των κρατών που απειλούν τις επενδύσεις τους η Αυστραλία το 2005 αρνήθηκε τη ρήτρα αυτή ISDS, θεωρώντας ότι το νομικό του σύστημα ήταν αρκετά ισχυρό για να λύσει τέτοια προβλήματα. Άλλη ερώτηση. Τι πρόβλημα έχει λοιπόν το καναδικό ή το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα, ούτω ώστε να χρειάζεται το σύστημα ISDS. Πέμπτον, ποιες προϋποθέσεις ε, θα θέσουν οι επιχειρήσεις που θα ε, καταπατούν τα δημοκρατικά δικαιώματα των λαών και πώς θα επιβληθούν αυτά μέσω του ISDS. Τι είδου ε, ποσά θα ζητηθούν σε αποζημίωση και πώς έτσι μια επιχείρηση μπορεί να ε, επηρεάσει ένα δημοκρατικό κράτος. Το πόσιμο νερό. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν μια πρωτοβουλία πολιτών για να παραμείνει δημόσιο αγαθό το νερό. Η Κομισιόν τι κάνει για να εξασφαλίσει ότι το πόσιμο νερό δεν θα γίνει ε, μείνει, ε, στο έλεος της, δημόσιας, της ε, ιδιωτικής αγοράς. Ε, πρόσφατα στην Ολλανδία χαρακτηρίστηκε η χώρα φορολογικός παράδεισος. Φαντάζομαι ότι ξέρω τι εννοείται. Η τελευταία μου λοιπόν ερώτηση είναι έχει δει κανεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα ενός φιλικού φορολογικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με το ISDS. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Κάποιες από τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω έγιναν ήδη από άλλους για το ISDS. Ακούσαμε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει εντολή διαπραγμάτευσης αλλά η συμφωνία με τον Καναδά μας είπαν ότι θα είναι βάση για τη διαπραγμάτευση για τη Διατλαντική Συμφωνία. Μας είπαν ότι βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα, η διαδικασία όμως έχει ολοκληρωθεί και δεν μπορούμε να επανέλθουμε. Δηλαδή μας καλείται σήμερα να κυρώσουμε μια αμφισβητούμενη διαδικασία και να δημιουργηθεί έτσι ένα τετελεσμένο γεγονός, μια νομολογία και μας λέτε ότι δεν μπορούμε να οπισθοχωρήσουμε. Και βεβαίως όταν ολοκληρωθεί και η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας πείτε το ίδιο. Αφού ολοκληρώθηκε η Συμφωνία του Καναδά δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα δημοκρατικό θέμα, θέμα δημοκρατικής νομισμότητας και γι' αυτό και εκφράζονται αυτές οι ανησυχίες όσον αφορά την ενδεχόμενη κύρωση της συμφωνίας. Δεύτερο σημείο, οι, μη, ε, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Υπάρχει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό και η διαμάχη και το αρμόδιο όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ έχει εκφραστεί. Η Ευρώπη λοιπόν είπε ότι δεν θα επιβάλλει κάτι παραπάνω στον Καναδά. Ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούνκερ, στην προεκλογική του εκστρατεία και στις ακροάσεις του, είπε ότι επιθυμεί να βελτιωθεί η αξιολόγηση και η αδειοδότηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στην Ευρώπη. Αν λοιπόν βελτιωθεί η αξιολόγηση αυτών των οργανισμών στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τον αντίκτυπο στην υγεία κτλ. Τι θα κάνει ο Καναδάς σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, αν λάβει χώρα. Τρίτον, στο, για το SPS δεν είδα πουθενά κανένα μέτρο που να αφορά την υγιεινή Παραδείγματο χάρη. Στο παράρτημα Β υπάρχει καταρχήν παράρτημα Β και μπορούμε να το εξετάσουμε. Το παράρτημα Β θα προετοιμαστεί αργότερα. Θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το περιεχόμενό του. Για τα γενώσιμα, τέλος, έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση του Καναδά όσον αφορά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στο τομέα της υγείας για το επιπλέον κόστος, ιδιαίτερα για την πρόσβαση για κάποια ειδικά φάρμακα. Τέλος, αναφερθήκατε στην βιώσιμη ανάπτυξη, πολύ θετικό αυτό. Και βλέπουμε και στην Διατλαντική Συμφωνία ότι η Ευρώπη είναι πολύ πολύ διστακτική όσον αφορά το δεσμευτικό χαρακτήρα ενός τέτοιου κεφαλαίου. Πώς του εξηγείται αυτό, γιατί είναι τόσο μα τόσο επιφυλακτική η Ευρώπη για τα θέματα αυτά και απλώς τα αναφέρει επικοινωνιακά. Ευχαριστώ πολύ φιλελεύθερη. Τελικά κάποιος να πάρει το λόγο από τους φιλελεύθερους. Όχι. Ο κύριος Σούστερ. ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος, παραδείγματος χάρη. Ο Καναδάς δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιώτο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ να υπάρξει κάποια αντίφαση. Υπογράφουμε δηλαδή με τον Καναδά, ενώ ε, υπάρχουν άλλες ε, περιβαλλοντολογικές προβλέψεις από μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπόρεσα να ελέγξω τίποτα, αφού δεν έχουμε ακόμα το κείμενο της συμφωνίας. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, και εδώ υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2011 τον Νοέμβριο είναι πολύ συγκεκριμένη για το θέμα του ISDS. Η Επιτροπή λοιπόν λαμβάνει υπόψη του αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση, είναι πολιτικό θέμα και αν πρέπει να κυρωθεί η συμφωνία πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, δεν είναι δυνατόν το ISDS να συμπεριληφθεί χωρίς καμία εξέταση σε αυτό το κείμενο. Η συμφωνία αυτή η οικονομική εταιρική σχέση με τον Καναδά συμπεριλαμβάνει αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι και των δύο συμφωνιών η κύρωση δεν μπορεί να γίνει χωρίς ανοιχτά να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Και δεν μπορεί να μας αγνοεί η Επιτροπή και να κάνει ό,τι θέλει. Είτε λοιπόν θα βγει το θέμα αυτό από την συμφωνία, είτε θα αναβληθεί η κύρωση. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που έχει κοινωνικές πολιτικές επιπτώσεις. Πρέπει εμείς να μπορούμε να δικαιολογήσουμε γιατί αυτό το κείμενο έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία. Είτε λοιπόν θα βγει από το κείμενο, είτε θα πρέπει να αναβληθεί η κύρωση. Σε δύο εβδομάδες δεν θα είμαστε σε θέση στο Στρασβούργο να πάρουμε απόφαση και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε πρόκειται για μια καλή συμφωνία. Ό,τι λοιπόν συμπεριλαμβάνει είναι καλό. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι η ΣΥΤΑ είναι μια συμφωνία ιστορική ε, διμερής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια άλλη προχωρημένη, ε, ανεπτυγμένη οικονομία του ΩΣΑ. Συνεπώς ε, πρέπει ε, να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε ορισμένα θέματα. Και υπάρχουν δύο σημεία που θέλω να αναφέρω. Ένα αναφέρθηκε από τον David στα σχόλιά του σχετικά με το κεφάλαιο αηφόρου ανάπτυξης. Νομίζω ότι υπήρξε μια χαμένη ευκαιρία ε, να έχουμε ένα καλό κεφάλαιο για την εργασία. Είναι μια διαφορετική βεβαίως συζήτηση για το περιβαλλοντικό ε, κεφάλαιο ε, υπάρχει ε, δύο χωριστά κεφάλαια, ένα για την εργασία, ένα για το, το περιβάλλον και είναι λυπηρό που κανένα από αυτά τα κεφάλαια δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι σε σχέση με τις συμφωνίες που συνάψαμε με άλλες χώρες, η εφαρμογή της εποπτείας, της παρακολούθησης, χωρίς καμία αναφορά σε πρότυπα δεσμευτικά ε, δεν είμαστε μια συμφωνία ναύτα πλάσα ε, ε, που συνήφθη πριν από 20 χρόνια. Αυτό είναι το ένα σημείο και θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει η Κομισιό ποια, ποια είναι η λογική σύμφωνα με την οποία είναι καλό αυτό το κεφάλαιο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι υπάρχουν ε, μερικά καινοτομίε ή εξελίξεις σε σχέση με τη ΣΥΤΑ, πρώτα απ' όλα το πεδίο ε, εφαρμογής και επίση η μεγάλη απολευθέρωση των υπηρεσιών στην ε, συμφωνία. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται μια τέτοια συμφωνία. Έχουμε επίσης μια, ένα τέτοιο κατάλογο αρνητικό θα ήθελα να κάνω έκκληση στην Επιτροπή, διότι η διαφάνεια δεν είναι μόνο η δημοσίευση ε, εγγράφων, αλλά θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι σημαίνουν αυτά τα έγγραφα, τα κείμενα, να ξέρουμε πολύ καλά τι περιλαμβάνεται ε, στις υπηρεσίες, ε, στις υποχρεώσεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες γίνονται ένα μεγάλο πολιτικό θέμα παντού και νομίζω ότι είναι ουσιώδες να έχουμε διαφάνεια στο θέμα αυτό. Αυτά είναι τα δύο σημεία για τα οποία περιμένω μια απάντηση από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ στην Επιτροπή που μας έδωσε εξηγήσεις. Μικρόφωνο ε, τις εξηγήσει ε, που μας έδωσε σήμερα για το θέμα. Σχετικά με την Επιτροπή αναγνωρίζεται ότι η Συμφωνία Επιτάπητος δεν είναι ευθυγραμμισμένη με την τελευταία συζήτηση που είχαμε. Είναι μια ομολογία από την Επιτροπή ότι δηλαδή σήμερα υπάρχουν συζητήσεις πολιτικές αλλά δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε την ατζέντα που είχαμε και έχουμε ένα κείμενο που δεν λαμβάνει υπόψη την πολιτική συζήτηση. Ευχαριστώ που το αναγνωρίζετε ε, και υπενθυμίζω τα όσα μας είπε ο κύριος Γιούνκερ πριν από τις διακοπές και που λέει δεν θα δεχθώ η δικαιοδοσία των δικαστηρίων των κρατών μελών να περιορίζεται από ειδικά συστήματα σχετικά με τις ε, διαφορές, τη διευθέτηση των διαφορών ανάμεσα σε επενδυτές και κράτος. Νομίζω ότι το κείμενο ε, το οποίο μας υποβλήθηκε τώρα δεν είναι σύμφωνο με την δήλωση την πολιτική του σημερινού Προέδρου της Επιτροπής. Θα βρεθούμε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση όπου σε μια σύνοδο κορυφής Ευρώπης-Καναδά θα υπάρχει μια, θα υπογραφεί μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι σύμφωνη δεν ξέρω με το Συμβούλιο, αλλά με την νέα Επιτροπή το πρώτο θέμα λοιπόν που θέτω και νομίζω ότι ήδη ε, αναφέρθηκε σε αυτό το πλαίσιο το μεταβατικό, το πολιτικό, δεν θα ήταν καλύτερη επιλογή εκ μέρους της Επιτροπής να αναβάλει την υπογραφή, την μονογράφηση αυτής της συμφωνίας. Η μονογράφηση βεβαίως είναι μονογράφηση, αλλά όταν μονογραφηθεί ένα κείμενο απλώς υπάρχουν διαδικασίες, διατυπώσεις και δεν υπάρχουν πλέον ε, δυνατότητες ε, μεταβολών πολιτικών. Θα πούμε ναι ή όχι, είναι αυτοκτονία εκ μέρου της Επιτροπής να προχωρήσει με μια τέτοια συμφωνία, διότι θα έχουμε κρίση στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να επικυρώσει, να υπογράψει, να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία, αλλά θα υπάρξει και το στάδιο των κρατών μελών ε, που θα πρέπει επίσης ε, να αποφανθούν. Κάποιος είπε ότι χρειάστηκε χρόνος για τις διαπραγματεύσεις, ένας μήνας λιγότερος, ένας μήνας λιγότερο, δεν θα αλλάξει τίποτα στις σχέσεις μας, τις οικονομικές με τον Καναδά. Το άλλο το θέμα είναι το θέμα ε, της ε, χρήσης για πρώτη φορά των αρνητικών καταλόγων που είναι επικίνδυνοι. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε αρνητικούς καταλόγους που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο διότι είναι σαν να λέμε όλα είναι εφικτά εκτός από. Αλλά όταν λέμε όλα είναι εφικτά εκτός, εάν ε, δεν έχουμε διευκρινίσει σαφώς τα πράγματα, ό,τι δεν έχει διευκρινιστεί σαφώς είναι θέμα απελευθέρωσης και βρισκόμαστε με ένα διακύβευμα με μίσα που κινδυνεύουν να έχουν απελευθέρωση, που είναι τεράστιος κίνδυνος. Εγώ προτιμώ τους θετικούς καταλόγους και όχι τους αρνητικούς. Τρίτο σημείο, είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Διάβασα στην συμφωνία ότι ο Καναδάς θέλει να προστατεύσει όλες, όλους τους πολιτιστικούς κλάδους και βιομηχανίες, ενώ η Ευρώπη προστατεύει μόνο τον οπτικο-ακουστικό τομέα. Γιατί αυτή η διαφορά, η διάκριση, γιατί η Ευρώπη δεν προστατεύει περισσότερο την κουλτούρα, τον πολιτισμό, εμείς προστατεύουμε λιγότερο την πολυμορφία μας, την πολιτιστική. Από ό,τι άκουσα συζητήσει για το TTIP, το Διατλαντική Εταιρική Συμφωνία, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η στάση της Ευρώπης σε σχέση με αυτήν την ιδιαιτερότητα των οπτικοακουστικών και όχι της κουλτούρας, του πολιτισμού γενικά. Και το τελευταίο σημείο αναφέρεται ε, στο ό,τι λένε οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που λένε ότι προστατεύουμε τα πρότυπα όπως έχουν σήμερα που δεν μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε πρότυπα γενικού συμφέροντος που θα μπορούσαν να προστατεύσουν για το μέλλον. Τι περιθώριο δίνει στον εαυτό της η Ευρώπη για να διαπραγματευτεί ανώτερα πρότυπα για την προστασία των πολιτών της προς το γενικό συμφέρον. Ποιο είναι αυτό το περιθώριο ελιγμού που ενέχεται σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Άλλοι τρει έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ολοκληρώσουμε με τι ερωτήσει και κατόπιν θα πάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ενδιαφέρον τη συζήτηση και ιδιαίτερα την παρουσίαση του κυρίου και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι γιατί ως μέλος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά στο προηγούμενο κοινοβούλιο ε, συμμετείχα στις ε, συζητήσεις αυτές και ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ε, πρόθεσαν την υπόθεση αυτή. Μπορώ να δω γιατί είναι τόσο ενθουσιώδης ο κύριος Πατριτσιών για τα όσα επιτεύχθησαν. Ε, χρησιμοποιεί εκφράσεις ε, όπως εκπληκτικό αποτέλεσμα, ε, πρωτοπόρες λύσεις κλπ. Αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ε, βέβαια. Ελπίζω ότι η συμφωνία αυτή θα έχει επιτυχία, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα σχετίζεται με τη διαδικασία. Είπε ότι θα κυκλοφορήσει το κείμενο στις επαρχίες του Καναδά. Πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι επαρχίες ή είναι μόνο για διαβούλευση ε, που θα κυκλοφορήσει το κείμενο και θα αποφασίσει η εθνική κυβέρνηση τελικά. Δεύτερον, μια πιο ε, ε, συγκεκριμένη λεπτομέρεια σχετικά με την απελευθέρωση των δασμών στη Γεωργία που είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους γεωργούς μας και θέλουν να έχουν διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις. Και τρίτον, υπάρχει μια ρήτρα επανεξέτασης ούτως ώστε, ότι, ούτως ώστε αν κάτι δεν πάει σύμφωνα με τα σχεδιαζόμενα να μπορέσει να διορθωθεί. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα επανέλθω σε δύο σημεία Κάποια από τις προηγούμενες ομιλήτρες μίλησε για τις αρνητικές και τις θετικές λίστες και καταλόγους. Ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε υπέρ της ύπαρξης αρνητικών καταλόγων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά ε, τα θέματα, καθώς και η διάρκεια θέσης σε ισχύ κάποιων προθεσμιών, κάποιων κατηγοριών προϊόντων. Θέλουμε πραγματικά να προωθήσουμε την ανάπτυξη και θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε άλλες περιοχές του κόσμου με ευνοϊκές συνθήκες. Χρειάζεται λοιπόν, όπως ξέρετε, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, η μεγαλύτερη δυνατή, έτσι ώστε να δώσουμε κάποιες εγγύησεις και κάποια ασφάλεια. Όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων. Όλα όσα συζητούμε σήμερα δεν είναι προαποφασισμένα. Αυτό που σίγουρα μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια συμφωνία που να εγγυάται τα δικαιώματα ενός ξένου επενδυτή. Πώς ε, λοιπόν θα λύσουμε θέματα διαφάνειας, ε, εναλλακτικών δυνατοτήτων επένδυσης. Είμαστε στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων. Τα τελευταία τρία χρόνια αυτό κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και πραγματικά η έκθεση Καντέρα Ρίφ έχει ακριβώς αυτό το θέμα. Με μεγάλη σοβαρότητα συζητήσαμε όλες αυτές τις πτυχές του θέματος. Και θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να ξαναδούν αυτήν την έκθεση τι σημαίνει προστασία του επενδυτή σε άλλες χώρες όπως τον Καναδά και αλλού. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει πάνω από 2.000 συμφωνίες που περιλαμβάνουν προστασία του επενδυτή με χώρες όπως αυτές της Λατινικής Αμερικής και αλλού. Και εξηγήστε στους φτωχούς των χωρών αυτών ότι το σύστημα της χώρας τους δεν είναι τόσο ασφαλές όσο αυτό της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγήστε επίσης και στους Κινέζους ότι θέλετε να υπογράψετε συμφωνίες με τέτοιου είδους προδιαγραφές και πρότυπα, κάτι που ποτέ δεν πρόκειται να δεχτούν. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ εδώ σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντάς τους ότι από τη στιγμή που συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια, κάποια προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια των επενδύσεων και την προστασία των επενδύσεων. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες συμφωνίες της δεκαετίας του 60, του 70 και αργότερα, όπου όλα τα θέματα δεν έχουν λυθεί. Είναι ίσως μια ευκαιρία για μας όταν υπογράφουμε συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Καναδά, με τέτοιες χώρες, είναι μια ευκαιρία, μια τύχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία τέτοιας ποιότητας όπου πραγματικά η ασφάλεια και η προστασία των επενδύσεων είναι τέτοιου επίπεδου. Και πραγματικά αυτό που ζητήσαμε για, την, για τις ε, επενδύσεις και την προστασία των επενδύσεων ελπίζω η Επιτροπή να το έχει λάβει υπόψη της και ξέρετε πολύ καλά ότι όλες οι ευρωπαϊκές επενδύσεις ζητούν να ληφθεί υπόψη αυτή η προστασία των επενδύσεων σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου αυτό είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, ξέρετε όμως ότι η προστασία των επενδύσεων δεν αποτελεί ένα από τα σημαντικά επιχειρήματα για να επιλεγεί μια χώρα είτε επένδυση. Όπως παραδείγματο χάρη, αυτή ήταν η απάντηση που πήραμε για τη Βραζιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Οι κυρίες πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να μας εξηγήσετε πώς δίνετε το λόγο, γιατί πάνω από 34 ώρες τώρα ε, ζήτησα το λόγο, μου κάνετε μήνυμα ε, σήμα ότι το σημειώσατε, αλλά τι γίνεται, κάνα μία ερώτηση. Εκφράζω την πρώτη ομάδα των ε, Γάλλων ε, Ευρωβουλευτών. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ούτε η γραμματεία, ούτε εγώ το σημειώσαμε. Μήπως πρέπει να σκόνετε λίγο πιο ψηλά το χέρι σας στο μέλλον. Εγώ θα... Ευχαρίστως να παραχωρήσω το λόγο και να επανέλθω μετά, λέει ο κύριος quel dirigisme on aurait pu parler l'un et l'autre mais c'est vrai que ça aurait probablement été deux voix de critique. Ναι, ναι, βεβαίως ξέρω ότι η Κομισιόν δεν της αρέσουν οι κριτικές, οι αμφισβητήσεις, αυτό που βλέπω ότι η αλήθεια αναδύεται ευκολότερα μετά τις εκλογές από ό,τι πριν, διότι πριν από τις εκλογές είπαμε ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά θα είναι το πρόχειρο έγγραφο για να αντιγραφεί μετά από την Διατλαντική Συμφωνία εταιρική Σχέσης. Μας είπαν όχι, όχι δεν είναι έτσι μετά τις εκλογές, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αλήθεια. Βεβαίως αυτή η συμφωνία, αυτό το κείμενο βεβαίως θεσπίζει μια ιδιωτική δικαιοσύνη ανάμεσα στις πολυεθνικές και τα κράτη και όχι μια δημόσια δικαιοσύνη μεταξύ επενδυτών και κράτους. Θα επιτρέψετε τους Γάλλους να είναι πάρα πολύ επικριτικοί απέναντι στα διαιτητικά δικαστήρια, αλλά μια φορά όπου χρησιμοποιήθηκε η λύση αυτή οδήγησε στην ανάκριση του αφεντικού του Διεθνούς νομισματικού ταμείου. Βλέπουμε πολυεθνικές στη Γαλλία θα θεωρήσουν ότι είναι, είναι οι κανόνες, δεν ευνοούν την, ε, ε, δική τους ε, δραστηριότητα και ότι το κράτος θα πρέπει όμως τότε να λάβει υπόψη το συμφέρον των πολυεθνικών προτού λάβει μια απόφαση. Η καναδική κυβέρνηση θα, απο, θα αποφασίσει ας πούμε το δικαιοστάσιο για το σχιστολιθικό πετρέλαιο όταν ζητήσει μια επιχείρηση 250 εκατομμύρια αποζημίωση όταν σκεφτεί ότι μια τέτοια διακοπή, ε, τότε τι έγινε, τι γίνεται με τους κανόνες της ναύτα. Ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι, εκατομμύρια Γάλλοι είναι ριζικά αντίθετοι στην ιδιωτική δικαιοσύνη, στην αδιάφανη χρησιμοποίηση τέτοιων μέσων και στην εξουσία των πολυεθνικών. Το μόνο θέμα που θα ήθελα να θέσω στην Επιτροπή είναι πότε ε, θα ε, τελειώσετε, θα μπορέσετε ε, να ακούσετε την άρνηση των λαών. Και ο τελευταίος last but not least. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη που άργησα, αλλά μιλούσα με δύο ψηφοφόρους μου που ήταν εδώ και η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι να ζητήσω διευκρίνηση από την Κομισιόν σχετικά με το timing, το χρονοδιάγραμμα, πώς μοιάζει να διαμορφώνεται για τη συμφωνία αυτή, ώστε να ε, επικυρωθεί και να τεθεί σε, ισχύ αυτή η συμφωνία, γιατί οι ψηφοφόροι μου ε, ανησυχούν πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, η κυρία Μαρία Ρένα, η σοσιαλίστρια ε, βουλευτής, είπε να έχουμε... Ε, να κάνουμε μια παύση στη συμφωνία με τον Καναδά αλλά οι ίδιοι στη σοσιαλιστική ομάδα ψήφισαν να επιταχυνθεί μια πολύ πιο αμφιλεγόμενη και εμπριστική ε, συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Ε, μπορεί κάποιος από τους σοσιαλιστές να μου εξηγήσει πού βρίσκεται η συνέπεια ανάμεσα στο να ζητάνε καθυστέρηση της συμφωνίας ε, με τον Καναδά που τώρα τη συζητάμε εδώ και τρία χρόνια τουλάχιστον ενώ ταυτόχρονα θέλετε fast track για αυτή την πραγματικά εμπριστική και ανησυχητική ε, συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία που είναι σχεδόν άνευ προηγουμένου. Θα μπορούσατε παρακαλώ να με διαφωτίσετε. Ίσως διμερώς θα σας διαφωτίσουμε, έτσι και θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ε, απόψεων αλλά και ερωτήσεων. Ίσως ε, μπορείτε να απαντήσετε κάπως ομαδικά. Καλή τύχη σας εύχομαι. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, τελικά θα δυσαρεστήσω πολλούς αν δεν καταφέρω να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Τώρα, όσον αφορά τις εξηγήσει σε μια συνεδρίαση σαν και αυτή, πολύ περιορισμένο χρόνο, κάτι το οποίο θα μου οδηγήσει ίσως μη ικανοποιητικές απαντήσεις. Με μεγάλη χαρά θα δώσω είτε στα μέλη της Επιτροπής είτε στους ε, βοηθούς τους πολύ πιο εμπεριστατωμένες απαντήσεις για τεχνικά θέματα. Όπως σας είπα, οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν 3 η ώρα το πρωί την 1η Αυγούστου. Και φυσικά θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξηγήσουμε σε όλους που ενδιαφέρονται για όλες τις λεπτομέρειες αυτής της διαπραγμάτευσης, κυρίως στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική εκτίμηση, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό θα το κάνει πολύ καλύτερα από μένα ο Επίτροπος. Και φυσικά εδώ δεν είναι και η τελευταία φορά που συζητούμε το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να σας δώσω όσο πιο πολλά στοιχεία συγκεκριμένα μπορώ και πληροφορίες που αφορούν αυτό το θέμα. Ξεκινώ τώρα με τα τρόφιμα, το βοιοκρέας. Ναι, έχετε δίκιο όσον αφορά τα πρότυπα. Η συμφωνία αυτή δεν εναρμονίζει, δεν αλλάζει τίποτα που αφορά το περιβάλλον, την υγεία, την δημόσια ασφάλεια και τα πρότυπα που θέτουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο θέμα, καθότι ο Καναδάς έχει παρόμοιες ανησυχίες με μας. Αναφερθήκατε στο βόλιο κρέας και την παραγωγή του Καναδά που συμπεριλαμβάνει ορμόνες. Ναι, έχετε δίκιο. Σε κάποια σημεία διαφέρουν τα πρότυπά μας. Μυστήστε όμως ότι είχαμε πολύ πιο περίπλοκες ε, περιπτώσεις και βρέθηκε λύση και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί λύση και για το βόλιο κρέας από τον Καναδά Μέχρι τώρα δεν έχουμε ανοίξει τον τομέα αυτό και φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένες ποσοστώσεις 0,6% της ευρωπαϊκής αγοράς μόνο για τα προϊόντα αυτά και δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τις δικές μας προδιαγραφές και πρότυπα για την εκτροφή και τον σφαγισμό των ζώων. Ζητούμε βεβαίως βόλιο κρέας χωρίς ορμόνες και ίχνη λασιμότητα και ασφάλεια και πιστοποίηση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν αλλάξαμε τίποτα λοιπόν όσον αφορά τους ε, εκτροφείς. Αναφερόμαστε εδώ για μια ποσότητα 46.000 τόνων και βεβαίως εδώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη ε, αλυσίδα εκτροφής και παρακολούθησης. Όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς τώρα. Αυτό που αναφέρθηκε και ο κύριος Ζαντό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ενσωματώσει στην συμφωνία. Υπήρξε ο ίδιος διάλογος, τον συμφωνήσαμε στην Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Μπορείου είναι κάτι που δεν εγγυάται τίποτα στον Καναδά. Όσον αφορά την εξέλιξη των ρυθμίσεων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς προϋποθέτει την εφαρμογή των ε, κανονισμών και ρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ τίποτα καινούριο. Μας πήρε πολλά χρόνια να πάρουμε απόφαση για το θέμα αυτό, για τη συμφωνία με τον Καναδά και αν ο Καναδάς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είχε άκαμπτη θέση, φυσικά δεν θα είχαμε φτάσει στο αποτέλεσμα που φτάσαμε. Και ρυθμίστηκαν τα επίμαχα θέματα, είτε αν θέλετε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε σήμερα, τα θέματα που έχουν ρυθμιστεί μετά από διαπραγμάτευση είναι αυτά που είναι και δεν θα τα ξαναδιαπραγματευτούμε. Θέλω επίσης να σας πω ότι όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Συμφωνίας του Καναδά και αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχω απολύτως ε, τίποτα να ε, απολογηθώ ή να διευκρινίσω και ίσως παρερμηνέθηκαν τα λόγια μου. Εγώ θα σας παρουσιάζω εδώ πολύ συγκεκριμένα ποια είναι η εντολή μας και ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν μεταξύ κοινοβουλίων, μεταξύ μελών της Επιτροπής, μεταξύ των μελών της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορώ λοιπόν να σας εγγυηθώ καμία εξέλιξη στο μέλλον συγκεκριμένη και δεν μπορώ να δεσμευθώ. Μπορώ να σας πω απλώς ότι το κείμενο αυτό δίνει απαντήσεις με ένα ισορροπημένο κατά την άποψή μας τρόπο, προστατεύοντας τα συμφέροντα των επενδυτών και διατηρώντας τη δυνατότητά μας να τηρήσουμε την νομοθεσία μας. Και αν συμφωνεί κάποιος ή όχι, είναι κάτι προσωπικό, είναι θέμα πολιτικής άποψης ή ιδεολογίας και δεν μπορώ εγώ εδώ να το επικρίνω. Στην ουσία, οι διαιτητικές διαδικασίες, όπως και οι δικαιοδοτικές ε, διαδικασίες στα δικαστήρια, αν θέλετε, ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν την νομοθεσία και προσπαθούν πάντα να λάβουν υπόψη τους τα συμφέροντα των δύο μερών. Όσον αφορά τις περιπτώσεις επενδύσεων, Όταν υπάρχουν παραδείγματο χάρη σαφείς υποθέσεις όπως απαλωτριώσεις, εκεί φυσικά υπάρχει η αποζημίωση. Αλλά σε καμία περίπτωση ένας επενδυτής δεν μπορεί να προσφύγει μόνο και μόνο για θέματα διαφυγόντος κέρδους. Και φυσικά μπορεί να προσφύγει μόνο όταν υπάρχει προφανής αδικία ή μέτρα τα οποία πραγματικά πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα ενός επενδυτή. Πρόκειται για μέτρα και για πρότυπα που εφαρμόζονται και λαμβάνονται υπόψη στην πάγια νομολογία αυτών των διαιτητικών δικαστηρίων και σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα αλλάξει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Γιατί χρειάζεται αυτή η διαιτησία, αυτή η διαιτητική διαδικασία. Γιατί τα εθνικά δικαστήρια βασίζονται στην εθνική νομοθεσία. Ένα δικαστήριο στον Καναδά θα εφαρμόσει την νομοθεσία του Καναδά και όχι τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έχουμε διαπραγματευτεί για αυτές τις οικονομικές σχέσεις με τον Καναδά. Έχουμε λοιπόν, αν θέλετε σήμερα, διαπραγματευτεί κάποιες προστασίες και εγγύησεις που δεν υπάρχουν στην νομοθεσία του Καναδά. Και υπάρχουν μέτρα, παραδείγματο χάρη απαλωτρίωσης, που απαγορεύουν πρόσβαση σε εθνικά δικαστήρια. Και εδώ μπορεί να υπάρχει παραδείγματο χάρη ένα νόμιμο δικαίωμα κάποιου να προσφύγει σε ένα δικαστήριο και η προστασία που του προσφέρει μια διαιτητική διαδικασία είναι σίγουρα υψηλότερη από αυτή. Έχουμε επίσης ε, διασφαλίσει διαφάνεια βάσει των ε, κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφάνεια στις διαιτητικές διαδικασίες. Και μπορέσαμε να έχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ καθησυχαστικά όσον αφορά τη διαφάνεια παραδείγματο χάρη και πραγματικά ναι μπορείτε να πείτε ότι είναι μυστική ειδικά ή μη διαφανή δικαστήρια, αλλά όχι σε αυτή την περίπτωση. Οι ουσιαστικοί κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται εδώ είναι κανόνες που λαμβάνουν υπόψη τους και το δημόσιο συμφέρον. Και σε καμία περίπτωση δεν ε, μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Όσον αφορά τώρα τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αλλά και θέματα φαρμάκων. Οι κανόνες που εδώ έχουν υιοθετηθεί και, διαπρα... και που... τους οποίους έχουμε διαπραγματευτεί για θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ισχύουν με δεσμευτικό τρόπο για τον Καναδά, στη συμφωνία με τον Καναδά, από τη στιγμή που ένα φάρμακο καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εδώ υπάρχει συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και αλλού, εάν ναι ή όχι, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ προϊόντων που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ε, προϊόντων που δεν καλύπτονται. Στην περίπτωση λοιπόν του Καναδά που αυτή η διάκριση επιβάλλεται με δεσμευτικό τρόπο και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα των γενώσιμων φαρμάκων. Έχουμε διαπραγματευτεί μια προστασία και όπως ξέρετε υπάρχει και μεγάλη ποσότητα γενώσιμων φαρμάκων που εξάγονται από τον Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη τώρα. Ε, δεν μπορώ να πω σε όλες τις λεπτομέρειες. Απλώς θα ήθελα να πω ότι με όλο το σεβασμό δεν συμφωνούμε ότι οι ουσιαστικοί κανόνες ε, στο κεφάλαιο αυτό είναι κατώτεροι από τους κανόνες της ναύτα. Είναι γεγονός ότι δεν είναι ένα ε, ενιαίο κεφάλαιο που έχουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ο Καναδάς όμως δεν έχει καθόλου κεφάλαιο. Έχει παράπλευρες συμφωνίες ξεχωριστές. Εμείς έχουμε ένα τίτλο με δύο τμήματα για την εργασία και για το περιβάλλον, αλλά έχουμε κοινού κανόνες, κοινά στοιχεία πολύ πιο παρόμοια με τη δική μας ε, προσέγγιση πιστεύουμε ότι έχουμε διασώσει την ουσία της ολοκληρωμένης μας προσέγγισης. Μεγάλη διαφορά στο θέμα των κυρώσεων για το κεφάλαιο που αφορά την εργασία. Ξέρω ότι γίνεται μια συζήτηση και εδώ ε, για το κατά πόσο θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μέχρι τώρα δεν είναι αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι οι κυρώσεις δεν είναι το κατάλληλο μέτρο για την αηφόρο ανάπτυξη και η λύση είναι η συνεργασία. Μπορεί να αλλάξουμε θέση σαν αποτέλεσμα της ε, συζήτησης που ανέφερα. Αλλά προς το παρόν η Κομισιόν πρέπει να παραμείνει πιστή στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν, όπως ξέρετε, καλά επιχειρήματα που λένε ότι ακόμα και οι ε, οικονομικές ε, κυρώσεις των ΗΠΑ που γίνονται με καλή πρόθεση δεν είναι αναγκαστικά οι κατάλληλες. Δεν θέλω να προδικάσω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά σας λέω πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Τώρα, ένα ιδιαίτερο θέμα που είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρει πολλά μέλη και όχι μόνο αυτά που κατάγονται από τη Σκοτία τα νομικά συμβούλια. Legal boards. Ε, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Ο Καναδάς από την αρχή δεν ήθελε να δεχτεί να καταργηθούν ε, ε, τα επαρχιακά μονοπόλια. Ούτε θέλαμε να έχουμε ε, τέτοια επεμβατικότητα. Από την άλλη μεριά, για το δικό μας εμπορικό συμφέρον δεν είναι δεκτά τα legal boards. Τώρα αλλάζουμε τους κανόνες και είναι πολύ τεχνικό αυτό το θέμα. Ε, μιλάω πάντως για το τέλος που οι ξένοι επενδυτές πρέπει να καταβάλουν για να επωφεληθούν από μια πρόσβαση σε ένα μονοπόλιο. Το τέλος αυτό θα υπολογίζεται από εδώ και πέρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση θα έχουμε και μια ρήτρα που θα αφορά τις αντιμονοπολιακές συμπεριφορές ε, των επενδυτών έξω από την δικαιοδοσία των επαρχιών. Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται αυτό σε αγορές τρίτων χωρών. Έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων που έχουν δώσει τον εαυτό τους ε, οι Καναδοί από τους κανόνες αυτούς και από το status quo. Αλλά τελικά... Ε, χωρίς να καταργούμε τα μονοπόλια που δεν ήταν στις προθέσεις μας, ε, έχουμε μια καλή συμφωνία. Ε, στο παρελθόν, μια δυναμία των συμφωνιών αυτών ήταν δεν υπήρχε ένα αποτελεσματικό τρόπο επίλυση των διαφορών. Αυτό τώρα το συμπεριλάβαμε στη συμφωνία μετά από ε, μακρόχρονες διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι είναι θετικές οι αντιδράσεις από αυτή την άποψη. Ε, ζητώ συγγνώμη, ακολουθώ την ε, σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις και γι' αυτό είναι κάπως συγκεχημένες οι απαντήσεις μου. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα διδάγματα που έχουμε ε, πάρει μέχρι τώρα. Ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο πολλά θέματα που μας πήραν δύο χρόνια για να λύσουμε με τον Καναδά θα ήταν ζητήματα που δεν έχουν οικονομική σημασία. Ταυτόχρονα έχουμε ένα πλήρες σύστημα ε, εμπορικών, ε, εμπορικής νομοθεσίας και το ίδιο έχει ο Καναδάς που δεν είναι ταυτόσιμα τα συστήματα αυτά και έπρεπε να γίνουν συμβατά. Αν είχαν οικονομικές συνέπειες ή όχι αυτές οι διαφορές αυτό δεν είχε σημασία. Ο νόμος θα έπρεπε, πρέπει να εφαρμοστεί ε, Εξίσου, είτε υπάρχουν οικονομικές συνέπειες, είτε όχι. Οι κανόνες προέλευσης ήταν ένα θέμα όπου οι διαπραγματεύσεις ήταν οι πιο δύσκολες που είχαμε μέχρι τώρα με οποιαδήποτε χώρα. Ε, έπρεπε όμως να ρυθμιστεί και το θέμα αυτό και χρειάστηκε πολύς χρόνος. Ο Καναδάς έχει ένα πολύπλοκο μηχανισμό λήψης αποφάσεων που συμπεριλαμβάνει και τις επαρχίες. Πρέπει να πω ότι οι επαρχίε που μα έδωσαν καταρχά πολιτικέ διαβεβαιώσεις ότι θα συμμετείχαν καλή την πίστη και αν ήταν ικανοποιημένε με το αποτέλεσμα θα εφάρμοζαν τη συμφωνία καλή την πίστη, έπαιξαν ένα πολύ επικοδομητικό ρόλο σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Αλλά βέβαια αυτό προσέθεσε στην πολυπλοκότητα της τη υπόθεση. Σύμφωνα με τη συνθήκη, έχουμε κι εμεί ένα πολύπλοκο μηχανισμό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα για να λαμβάνεται υπόψη η, πολυ... η ποικιλομορφία των κρατών μελών. Το ίδιο ισχύει και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Και αυτό δοκιμάστηκε τα τελευταία ε, έξι χρόνια. Ο Καναδάς προσπάθησε να επινοήσει ένα σύστημα συμμετοχής των επαρχιών του στις διαπραγματεύσεις αυτές για το διεθνέ εμπόριο. Έκαναν πολύ καλή δουλειά, αλλά αυτό πρόσθεσε στην πολυπλοκότητα του εγχειρήματο. Τώρα, τι θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου απλούστατα θα γίνει μια ανακοίνωση ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η κρίση της Κομισιόν. Σύμφωνα με όσα καταλαβαίνει η Κομισιόν, ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις και θεωρήσαμε ότι το να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση σε, α, σε ένα α ή σημείο δεν θα οδηγούσε σε περαιτέρω βελτιώσεις. Ολοκληρώνονται λοιπόν οι διαπραγματεύσει κατά την κρίση της Κομισιόν ω θεσμικού οργάνου. Λυπάμαι, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν θα ζητηθεί να ε, ε, εγκρίνει το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο για πολλούς μήνες ακόμα. Ε, ρώτησε κάποιος ποια είναι η το κοινοβουλιο για πολλους μηνες ακομα ε ρωτησε καποιο ποια ειναι η προβλεψη για το χρονοδιάγραμμα και την τελική κατάληξη. Δεν είναι δυνατό να κάνω τέτοια πρόβλεψη, αλλά δεν περιμένουμε τη θέση σε ισχύ πριν από το 2016, ίσως και αργότερα. Εξαρτάται πόσο καιρό θα χρειαστεί για την νομική ε, επανεξέταση, ε, για την νομική εξέταση μάλλον, για, την, ε, για τις μεταφράσεις, αλλά και για την πολιτική συζήτηση και εδώ και στον Καναδά. Δεν θα επιχειρήσω να κάνω μια πρόβλεψη για το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να γίνουν όλα αυτά. Πρόεδρε, Ξέρετε πάρα πολύ καλά ε, όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται ε, σχετικά με το αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέση σε ισχύ ή όχι. Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία αυτή από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Ε, δεν θα στοιχημάτιζα όμως σε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό με βάση την πείρα μου. Σας το λέω, δεν είναι η θέση του οργάνου που εκπροσωπώ. Τώρα, για το άλλο θέμα. Μιλάμε για μια ξένη χώρα εδώ. Από ό,τι ξέρω, οι επαρχίες δεν πρέπει επίσημα να εγκρίνουν τη συμφωνία. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να πρέπει να τροποποιήσουν την επαρχιακή νομοθεσία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Ο Καναδάς υποσχέθηκε ότι οι επαρχίες ακόμα και αν δεν πρέπει να εγκρίνουν την ε, συμφωνία, θα δώσουν την πολιτική τους ε, έγκριση και είτε θα τροποποιήσουν ανάλογα την επαρχιακή νομοθεσία ή θα εκδώσουν μια νομική πράξη που θα ε, δηλώνει ότι η νομοθεσία τους είναι συμβατή με τη συμφωνία. Επιμείναμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό από την αρχή της διαπραγμάτευσης. Η δημοσιότητα του κειμένου ο Καναδάς δεν ήταν πολύ, ήταν, τον απασχολούσαν, έπρεπε να επαναδιαγραφτεί με την ναύτα. Είναι, αν θέλετε, είναι δύο διαφορετικές συμφωνίες. Η δημοσιότητα, η δημοσιοποίηση του κειμένου. Αυτοί βεβαίως που κατακρίνουν έχουν δίκιο. Όπως είπα κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπε ο κύριος Ζαντό είναι ότι αυτό που διέρευσε είναι, δεν είναι οι απαντήσεις. Πάρα πολλά στοιχεία σημαντικά ε, λείπουν και έτσι δεν, μπορούσε κανείς, δεν μπορεί κανείς να κρίνει, κυρίως όσον αφορά τις υπηρεσίες. Με όλες τις επιφυλάξεις ακούω τις κριτικές για τον αρνητικό κατάλογο αν τον τρόπο με τον οποίο οι θετικοί ε, κατάλογοι ε, είναι γραμμένοι, δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά και πρέπει να δείτε πώς έχουμε γράψει ε, τις επιφυλάξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Θα δημοσιοποιηθούν και θα μπορέσετε να κρίνετε en connaissance de cause. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι δεν μπορεί κανείς να ζητάει κρίση από κάποιον χωρίς να έχει πλήρη γνώση του κειμένου. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι είναι το σωστό κείμενο. Και αυτό το κείμενο ακόμη και μετά από 27 ε, έτη πολιτικής εμπορικής δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντάξει κανείς ένα κείμενο. Θέλουμε όλα τα πράγματα να είναι σωστά. Θα είναι ένα νομικό έγγραφο. Είναι η Βεβαίως η συμφωνία έχει πάρα πολλές ρήτρες διατάξεις αναθεώρησης και θα μπορεί κανείς να κρίνει αν αυτό είναι απαραίτητο. Ακόμα πιο σημαντικό ε, είναι το θέμα των μελλοντικών κανονισμών. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Το δικαίωμα, ε, το κανονιστικό είναι προστατευμένο. Είτε οι κανόνες αυτοί καθεαυτοί είναι σαφώς ικανοί να αφήνουν περιθώριο ελιγμού, ώστε να αναπτύξουμε ε, κανονισμούς αντικειμενικούς που βασίζονται στα γεγονότα ή αν έχουμε αμφιβολίες για τα αν θέλουμε να αναπτύξουμε κανονισμούς στο μέλλον που για τον ένα ή άλλο λόγο ε, μπορεί να φαίνονται ή να είναι ε, να έχουν διακρίσεις, εκεί έχουμε επιφυλάξεις. Και πάλι δεν μπορείτε να κρίνετε μέχρι ότου να δείτε τα κείμενα. Δεν σας ζητώ λοιπόν ε, να ε, κρίνετε αυτά τα οποία λέω καλύτερα, ε, να δείτε τα κείμενα και να σας δώσουμε λεπτομερείς εξηγήσεις. Το θέμα των διαβουλέσεων για το TTIP. Ε, είναι για το TTIP και όχι για το ΣΥΤΑ. Εξετάζουμε τις απαντήσεις, δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε δεκάδες χιλιάδες απαντήσεις και επίσης ε, παρατηρήσαμε ότι μεταξύ 65-70 χιλιάδες ε, ήταν απαντήσεις στερεότυπες που προέρχονται από το διαδίκτυο. Μερικές δεκάδες χιλιάδες παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες γλωσσικές και υπάρχουν ακόμα χιλιάδες απαντήσεις που είναι πάρα πολύ λεπτομερείς, πολύ σημαντικές και χρειάζονται χρόνο ούτω ώστε και εμείς να μπορέσουμε να δώσουμε μια σοβαρή απάντηση. Αυτή η διαβούλευση αναφέρεται στο TTIP, η ΣΥΤΑ ε, δεν ξέρω τι είναι ένα κακό, μια κακή συμφωνία, δεν ξέρω, με βάση την εντολή που έχουμε αυτά κάνουμε για τον Καναδά. Και αν μας πείτε σταματήστε και να διαπραγματευτείτε ορισμένα τμήματα, αυτό θα είναι πολιτική απόφαση της Ένωσης, πολιτική απόφαση της Ένωσης. Και δεν μπορώ να κρίνω τι θα θέλει να κάνει το σώμα των επιτρόπων ή το μελλοντικό σώμα των επιτρόπων. Η δική μου άποψη, η άποψη η προσωπική μου είναι δεν ξέρω αν θα πρέπει να αναδιαπραγματευτούμε. Θα πρέπει τότε να αξιολογήσουμε τις συνέπειες. Αυτό που είπε η Επιτροπή μου για το TTIP είναι ότι ένα τέτοια, μια τέτοια, δεν είπα ότι είναι μεικτή συμφωνία και δεν νομίζω ότι είναι μεικτή συμφωνία. Εγώ νομίζω ότι ίσως το Συμβούλιο δεν συμφωνήσει μαζί μας. Αυτό συνέβη στο παρελθόν και το Συμβούλιο έχει την ε, κακή ε, τάση να προσπαθεί ε, να βρει ομοφωνία και ότι με τη μονοφωνία μπορεί να υπερισχύσει της Επιτροπής τέλος της ιστορίας τότε, αλλά αυτό θα συμβεί όταν παρουσιάσουμε την ε, συμφωνία για να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο. Ε, πόσιμο είδωρ, αν είναι ανθρώπινο δικαίωμα ή όχι, ε, δεν υπάρχει σε αυτήν την συμφωνία, σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, απελευθέρωση ε, του πόσιμου ύδατος. Έχουμε θέματα ε, για τα απόβλητα, για την διαχείριση των υδάτων. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να απελευθερωθεί. Νομίζω έχουμε επιφυλάξεις για αυτή τη θέση απέναντι στον Καναδά. Εξετάστε τις επιφυλάξεις όταν δημοσιοποιηθεί το κείμενο. Επίσης ο Καναδάς αναφέρει ένα θέμα ε, το, ε, η, προστασία του ύδατος τόσο ώστε να παραμείνει στην φυσική του κατάσταση. Ο Καναδάς έχει πάρα πολλά ύδατα τα οποία μοιράζεται με άλλες χώρες είναι σαφές ότι εμείς μπορούμε να δεχθούμε, να ικανοποιήσουμε ένα τέτοιο αίτημα να μοιράζεται εταιρείε, δεν ξέρω τι, τι σκέφτεται ε, η Ολλανδική κυβέρνηση για τους φορολογικούς παραδείσους, για τις εταιρείε μαϊμούδες. Δεν θέλουμε να υπάρχει forum shopping, δηλαδή να διαλέγει κανείς την καλύτερη δικαιοδοσία και το καλύτερο νομικό σύστημα αλλά έχουμε εξασφαλίσει να μην συμβαίνει αυτό. SPS ε, ε, υπάρχει μια εξήγηση την οποία δεν κατάλαβα ούτε κι εγώ ίδιος. Μόλις καταλάβω θα σας το δώσω. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει το παράρτημα Β ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει μελλοντικέ εξελίξει. Όταν καταλάβω εγώ ίδιος θα σας δώσω εξηγήσεις. Είμαι ο επικεφαλή διαπραγματευτή, αλλά δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του κειμένου αυτού. Επίσης ο συνάδελφός μου παρατηρεί ότι μερικοί από εσά είδατε το κείμενο των επιφυλάξων, διότι εστάλει στο Συμβούλιο που το κοινοποίησε ίσως το Κοινοβούλιο σύμφωνα με την συνήθη διαδικασία. Ίσως όλοι δεν έχουν πρόσβαση το θέμα του Καναδά σχετικά ε, με το περιβάλλον, ε, το κιότο, τα περιβαλλοντικά αγαθά. Υπάρχει διαφορετική στάση απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος. Ε, σύμφωνα με την πολιτική κατάσταση στον Καναδά υπάρχει συζήτηση, τα θέματα άλλαξαν στον Καναδά και θα αλλάξουν και άλλα. Έχουν περιπλακεί τα πράγματα, αλλά η συμφωνία δεν έχει να κάνει με το κιότο, ε, δεν ασχολείται με τα πράσινα προϊόντα και αγαθά. μιλάμε για πλήρη απελευθέρωση δασμολογική αντίθετα με τον πό και αυτά που αποκλείστηκαν ε, μιλάνε εκεί για πουλερικά και αυγά. Αυτά δεν θεωρούνται πράσινα ε, προϊόντα. Τα πράσινα προϊόντα και αγαθά ορίζονται αυτόματα. Ελπίζω να απήντησα σαφή εξήγηση ε, του τι είναι η επιφύλαξη ε, σχετικά με τις, ε, τις επιχειρήσεις κοινή ωφελία. Ξέρω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το νόημα αυτής της διάταξης. Δεν είχαμε συζήτηση με τα κράτη-μέλη και δεν εξετάσουμε ε, την ιδέα αυτή. Στο τέλος υπήρξε ε, μία σαφής άποψη ε, στην, στο Συμβούλιο για να έχουμε την ίδια γλώσσα με τον ΚΑΤ, ούτως ώστε να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία κάναμε δεν είχαμε νομική ανάλυση που να δείχνει ότι λειτουργεί εξίσου ε, καλά με την τον αρνητικό κατάλογο. Αν αυτό είναι η καλύτερη γλώσσα που μπορείτε να έχετε για να προστατεύσετε τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, νομίζω ότι ε, στο Συμβούλιο υπάρχει περίπου ομόφωνη γνώμη ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη γλώσσα. Πρέπει να πω βεβαίως ότι ο Καναδάς έχει διαφορετική άποψη έχουν διαφορετική άποψη, αλλά εμείς τους πείσαμε να ακολουθήσουν τη δική μας. Ε, σχετικά με την πολιτιστική βιομηχανία σε σχέση με την οπτικοακουστική. Αυτό είναι δύσκολη συζήτηση στο Συμβούλιο έχουμε την συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα οπτικοακουστικά αποκλείονται από την απελευθέρωση. Δεν βρίσκεται τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κονσένσου στο Συμβούλιο. Ο Καναδάς είναι διαφορετική χώρα, έχει διαφορετικές ανησυχίες, διαφορετικές βλέψεις. Αυτό που έχουμε στο ΣΥΤΑ δεν είναι η ε, προσέγγιση αυτή. Ε, ο Καναδάς αν ήθελε να αποκλείσει από τη συμφωνία όλα τα πολιτιστικά αγαθά θα μας έδινε διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν θα έχουμε την προστασία copyright ε, προς όφελος των συνθετών μας και των ε, συγγραφέων μας. Ποιοι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προστασία αυτή. Και έχουμε επενδύσεις στον Καναδά σε πολιτιστικό τομέα δεν δίνουμε τέτοιο δικαίωμα στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν επενδύσεις και όταν οι επενδυτές έχουν, δικαιούνται την ίδια προστασία αυτοί οι επενδυτές. Όσον αφορά την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούμε την στάση που είχε παραδοσιακά η Ένωση και έχω πλήρη επίγνωση ότι η θέση αυτή δεν εγκρίνεται πλήρως στην Ευρώπη, αλλά αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Επιτροπή δεν μπορεί να επινοήσει κάτι διαφορετικό σαν αφορά τον Καναδά. Έχουμε κάτι που προστατεύει τον Καναδά, ενώ συνάδει με τα δικά μας συμφέροντα. Ναι, η ερώτηση Κέλλη για τη γεωργία. Όπως είπα, αποκλείσαμε από τη συμφωνία την απελευθέρωση ε, για τις ε, χαλοπούλες, ε, τα πουλερικά, τα αυγά και έχουμε ποσοστώσεις για το βοδινό κρέας, το χοιρινό κρέας και για το τυρί, για τα γαλακτοκομικά. το μέγεθος των ποσοστώσεων δίνει στον Καναδά σημαντική πρόσβαση στην αγορά, αλλά εδώ η αγορά είναι περιορισμένη ανάμεσα στα κατεψυγμένα, στα νοπά και στην εδραίωση. 50.000 τόνοι βοήου συνολικά και 75.000 για το χοιρινό ε, και μπορώ να σας στείλω τον ε, λεπτομερή κατάλογο με μηδέν δασμούς αυτό σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά είναι μηδαμινές ποσότητες σημαντικές βεβαίως για τον Καναδά. Από τον Καναδά και δεν σας λέω τις τεχνικές λεπτομέρειες λάβαμε 18.500 για τυρί ε, που είναι ένα μικρό ποσοστό σύμφωνα με, την, ε, μερίδιο σύμφωνα με τον ΠΟΕ. Περιορισμένη πρόσβαση, αλλά λόγω των τιμών αυτών ε, των προϊόντων είναι κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο για τους εξαγωγείς μας και είμαστε ευτυχείς ε, που μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες ε, σχετικά με το θέμα αυτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Ελπίζω ότι απήντησα περίπου σε όλα. Ε, λυπούμε αν ξέχασα κάτι και πάλι για τις τεχνικές λεπτομέρειες θα είμαι διατεθειμένος να δώσω στο μέλη, στους βοηθούς τους τις εξηγήσεις που δεν θα βρείτε στο ίδιο το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Πάρα πολύ ολοκληρωμένη απάντηση. Ίσως αν κάποιοι θέλουν επιπλέον διευκρινήσεις, Σίγουρα αυτό θα μπορέσει να γίνει αργότερα, θα συνεχιστεί η συζήτησή μας. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση, διότι παρακολούθησα πάρα πολύ προσεκτικά αυτό που είπατε για την προσωρινή εφαρμογή, επειδή ακριβώς έχουμε προηγούμενο με την Νότια Κορέα, το Περού και την Κολομβία και η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει προηγουμένως να ε, εξετάσουν το κείμενο και να δοθεί η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το λέω με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και με αυτό το σημείο και πρέπει στο 17. Στα διάφορα δεν βλέπω τίποτα, άρα δεν θα εξετάσουμε κανένα σημείο. Και η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης θα λάβει χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου και θα ζητήσω από τους συντονιστές να παραμείνουν εδώ στην αίθουσα και όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να φύγουν.